Chers collègues, euh, bonjour. Je vous souhaite. On a l'impression de Λοιπόν, ε, φαίνεται σαν να είχαμε χωρίσει πριν από πολύ καιρό, αλλά ελπίζω ότι όλοι υποφεληθήκατε. Ασχέτως της χώρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, σε κρίση όπου πέρασε ο καθένας τις διακοπές του και έτσι μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε και πάλι τις εργασίες μας. Σχετικά με την υιοθέτηση της ημερησίας διάταξης έχω λάβει από τον εισηγητή μας κύριο Νταρντέν μία αίτηση να αναβάλουμε την ε, ψήφιση για το, την έκθεσή του στο σημείο 9 της ημερησίας διατάξεως ε, και ε, είμαι ε, σύμφωνη να μεταφέρουμε αυτή την, αυτή την έκθεση και άρα το σημείο 14 θα συζητηθεί τον Οκτώβριο ενώ θα μιλήσουμε τώρα για το 9 ε, και η ψηφοφορία θα γίνει τον Οκτώβριο διότι νομίζω ότι είναι βασικό να μπορέσουμε να καταρτήσουμε την στρατηγική του 2020 διότι οι εμπειρίες μας μας έχουν διδάξει ότι αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο συνεργαζόμαστε καλύτερα. Ας διαθέσουμε λοιπόν αυτό το χρόνο αν δεν υπάρχει κάποιος που αντιτίθεται σε αυτή την απόφαση. Ε, δεύτερον, web streaming, ε, σας ε, το υπενθυμίζω για να μην κάνετε πολλές γκριμάτσες όταν μιλάτε όσον αφορά το θέμα των ανακοινώσεων, το σημείο 2 όπου αναφέρεται εις τις νέες αρμοδιότητες και την απασχόληση. Άλλη ανακοίνωση αναφέρεται εις τον το, ΦΕΜ και ε, το, ε, στο ε, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου επ' αυτού και τις διατυπώσεις για να υπάρξει απλοποιημένη διαδικασία. Υπήρξε μία ανταλλαγή απόψεων επ' αυτού και δεν υπήρξε αντίρρηση στην υιοθέτηση χωρίς τροπολογίες και ε, γι' αυτό θα υπάρξει ένα ψήφισμα σχετικά με αυτό το ταμείο, το EMF ε, και ε, η Πολωνία μας ε, ενημέρωσαν ότι υπάρχει μία ε, μειονότητα που μπλοκάρει ε, αυτή την συζήτηση μπορεί όμως να αρθεί μετά τις εκλογές στο τέλος του μηνός στη Λετωνία και είναι βασικό να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε εις την ανανέωση χωρίς διαπραγματεύσεις αυτή της απλή πολλής ε, επεκτάσεως της ε, λειτουργίας αυτού του ταμείου όταν θα υπάρξει πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση του Ταμείου στα πλαίσια των ε, διαπραγματεύσεων για τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές θα τα ξαναπούμε αλλά ε, προτείνω προς το παρόν να διατηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που έχουμε και στη συνέχεια θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ε, σχετικά με την εξέλιξη της σημαντικής ομάδας που μας στηρίζει διότι θα μας εγκαταλείψει ε, ε, ο ένας συνάδελφός μας. Ε, λυπούμε πολύ, θα μας λείψει πολύ. Υπήρξε πάρα πολύ χρήσιμος και η εμπειρία του είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Τον ευχαριστώ και του είμαι ευγνώμων. Αλλά είμαι βέβαιη ότι ούτως ή άλλως αυτό θα γίνει σε κάποια εκδήλωση στις 12 του μηνός. Επίσης θέλω να χαιρετήσω και αναφέρω το όνομα για πρώτη φορά στη Σεβερίν Καγιά. Ε, σηκωθείτε. Είναι η πρώτη δοκιμασία να σας καλωσορίσουμε. Η ημερήσια διάταξή μας λοιπόν προβλέπει στο σημείο 3 την εξέταση των τροπολογιών σχετικά με το σχέδιο γνωμοδοτήσεώς μας για τον προϋπολογισμό του 2012, επί του οποίου είμαι εγώ εισηγήτρια και επί του οποίου θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Πρέπει όμως να βρω το φίλο μου. λοιπόν, σχετικά με τον προπολογισμό. Όπως πέρυσι έχουμε δύο έγγραφα και έχουμε δύο γνωμοδοτήσεις. Ένα που αναφέρεται εις ε, τις ε, δημοσιονομικές ε, προοπτικές ε, ε, και το άλλο ε, της ουσίας και ορισμένες τροπολογίες αναφέρονται σε ένα από τα δύο μόνο έγγραφα ενώ κανονικά θα πρέπει να, να υπάρξουν προτάσεις και για τα δύο δηλαδή και για τις ιδέες και για τους αριθμούς που, στους οποίους αναφέρονται. Υπάρχει λοιπόν μία, ε, ε, μία ε, τροπολογία του Έλμαρ και εγώ συμφωνώ με το σημείο αυτό. Πέραν αυτού όμως υπάρχουν τρεις τροπολογίες των πρασίνων σχετικά με ένα πολύ βασικό θέμα για τους απασχολείς των νέων και τα λοιπά και ε, στηρίζω. Δύο τροπολογίες της κυρίας Άρκιν ε, και οι άλλες ίσως ε, μειώνουν ε, τον ενθουσιασμό μου σχετικά με την αύξηση του, της χρηματοδοτήσεως του ταμείου επί του οποίου δεν θα συμφωνήσω γιατί γνωρίζετε τη γνώμη μου. Η, Υπάρχει ε, μια επιτροπή η οποία προτείνει να ε, διπλασιάσουμε την ε, την ε, χρηματοδότηση του Ταμείου ο, πρόκειται για τροπολογία της ΓΚΟΕ και ο κύριος Μπουρλό μας ζητά να στηρίξουμε ε, την ε, χρηματοδότηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες πρόταση που μπορούμε να στηρίξουμε στην επόμενη τροπολογία μας ζητούν να μην αυξήσουμε τις δικαιοδοσίες της ΕΚΤ και ε, ε, εγώ έχω κάνει μία τροπολογία σχετικά με τον προπολογισμό προόδου για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε το φόρουμ ε, και έτσι είχαμε χρηματοδοτήσει και το προηγούμενο. Και μια δεύτερη τροπολογία αναφέρεται σε την επέμβαση των επιθεωρητών εργασίας κατά των εταιριών που απλώς ε, είναι ε, ε, ένα γραφείο χωρίς ουσία για την επάνδρωση με εργάτες διαφόρων εργοταξίων. Έχω, έχω κάνει μία διερεύνηση αλλά δεν ξέρω που καταλήγει το θέμα αυτό. Επίσης θα πρέπει να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε ε, το σχέδιο προϋπολογισμού στις περικοπές που ζητά το Συμβούλιο αλλά ούσα μία πεπισμένη Ευρωπαία αλλά και ρεαλίστρια δεν μπορώ να στηρίξω τις προτάσεις αυξήσεως του προπολογισμού της Επιτροπής παρόλο που τις εύχομαι να επιτύχει. Όσον αφορά την κατάσταση στην Ελλάδα υπάρχει ε, μία συμφωνία που, στην οποία είχαμε καταλήξει εμείς ε, σχετικά με την έκθεση Κίνερ Πούντς και στην οποία δεν συμφωνεί το Συμβούλιο. Και τέλος ε, ε, πιστεύω ότι πρέπει να τροφοδοτηθούν οι σχετικές γραμμές. Σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία και την κοινωνική επανένταξη, όπως το κάνω και στην γνωμοδότηση, και εδώ προτείνω να συμπεριλάβουμε τη χρηματοδότηση του τέταρτου φόρουμ σε μια ε, τροπολογία που έχουμε συνυπογράψει με τον Φρεντερίκ Νταρντέν. Παρομοίω, ε, για, για την επιθεώρηση εργασία και του επιθεωρητέ εργασία, προτείνουμε την ενίσχυση ε, των σχετικών δημοσιονομικών γραμμών. Σε ό,τι αφορά τι τροπολογίε του ΕΛΚ τώρα, του συντονιστού μα του κυρίου Ρή, πολλοί ζήτησαν επαναφορά στα ποσά του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Χαίρομαι γιατί και εγώ αυτό πρότεινα αρχικά. Ενώ άλλες τοπολογίες ε, συστηματικά ζητούν αύξηση των ε, δαπανών, είτε των ε, λειτουργικών δαπανών, είτε των διοικητικών δαπανών. Και αυτό μου δημιουργεί πρόβλημα. Βλέποντας και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη συνειδητοποίηση της ανάγκης να έχουμε τη χρηματοδότηση των διαρθρωτικών ταμείων που θα συνοδεύεται από μια τεχνική αρρωγή. Αυτά είναι τα συμπεράσματα της 21ης Ιουλίου. Δεν τα συμμερίζομαι στο σύνολό τους, αλλά το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο επέμεινε στην ανάγκη η δέσμευση για τα διαρθρωτικά ταμεία ε, να συνοδεύεται από μια τεχνική αρρωγή και από μια εξακρίβωση της αποτελεσματικότητας της χρήσης των κονδυλίων. Εγώ πρότεινα να μην συμφωνήσουμε αυτές τις τροπολογίες του ΕΛΚ, όλο δε μάλλον που έρχονται σε αντίφαση με άλλες τροπολογίες του ίδιου μάλιστα του ΕΛΚ. Σε ό,τι αφορά τα πιλωτικά και πειραματικά προγράμματα, προτάθηκε να τροποποιηθούν οι σημειώσεις, οι παρατηρήσεις των συντονιστών και καταλήξαμε στη συμβαστική λύση και χαίρομαι γιατί το πιλωτικό πρόγραμμα για την ασφάλεια και την προστασία των εργαζομένων και του νέους θα παραμείνουν. Οι κύριοι Ορί και Κάστρες συνυπέγραψαν τέσσερις τροπολογίες. Ήταν ο εισηγητή μας για το, το ευρωπαϊκό έτος της γύρανσης και της δραστήρια γύρανση. Δύο τροπολογίες ζητούν την αύξηση των κονδυλίων για την επικοινωνία σε ό,τι αφορά την οργάνωση αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους δραστηρίας γύρασης, αγύρασης. Από τη μια λοιπόν το ΕΛΚ ζητά να καταργηθούν ορισμένες δημοσιονομικές γραμμές διοικητικών δαπανών και από την άλλη ζητά να αυξηθεί μία γραμμή επικοινωνίας. Ελπίζω το ΕΛΚ να αποσύρει αυτή την έκθεση, την ανθρωπολογία ή τουλάχιστον να την καταψηφίσουμε. Σε ό,τι αφορά το πιλωτικό πρόγραμμα την τροπολογία Μπουλό, που υπευλήθη σε άλλη επιτροπή για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ευρωμεσογειακή. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που ούτως ή άλλως εμπίπτει στις αρμοδιότητες της, ε, του οργανισμού ETF. Εγώ προτείνω προφορική τροπολογία στην τροπολογία ορή ώστε να έχουμε την ίδια τροπολογία για την ε, επανατροφοδίτηση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Κατάρτισης, του ETF, και θα σας διαβάσω την προφορική τροπολογία, μάλιστα την αρχική τροπολογία και την προφορική τροπολογία. Η αρχική τροπολογία προβλέπει ε, η προφοδοτή τον, ε, το Ίδρυμα αυτό με για την υποστηρίξη τις εταιρικές σχέσεις μεταξύ των μεσογειακών χωρών για την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και του συστήματος κατάρτισης καθώς και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου. Προτείνουμε προφορική τροπολογία στο τέλος αυτής της τροπολογίας και του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης, κόμμα, προώθηση του κοινωνικού διαλόγου και υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Αυτή είναι η προφορική τροπολογία, μια μικρή προσθήκη στην τροπολογία. Με τις τροπολογίες των πρασίνων συμφωνώ. Ζητούν την ενίσχυση της υποστήριξης προς τους νέους και τους κοινωνικούς εταίρους. Έχουμε δύο άλλες τροπολογίες της ΓΚΟΕ που προτείνουν αύξηση του προϋπολογισμού κατά τη γνώμη μου είναι η... εκτός πραγματικότητας αυτές οι τροπολογίες, γι' αυτό και δεν ε, τις υποστηρίζω προτείνω να τις καταψηφίσουμε. Περιμένω τώρα τα σχόλιά σας και τι θα γίνει με την προφορική τροπολογία για τη συμπερίληψη του, της τροπολογίας Μπουλόν. Ελπίζω να δώσετε το πράσινο φως και για αυτή την τροπολογία. Ποιος θέλει το λόγο παρακαλώ. Ο κύριος Σωρή και ο κύριος Σάρκας. Ευχαριστώ. Γενικώ συμφωνώ με όσα είπατε κυρία Πρόεδρε και θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις. για ορισμένα σημεία με τα οποία διαφωνώ. Το θέμα της αύξησης της μείωσης των προϋπολογισμών είναι ζήτημα επιλογής μάλλον. Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Ιουλίου ακολούθησαν τις δικές μας προτάσεις. Εμείς είχαμε καταθέσει τις τροπολογίες μας λίγο νωρίτερα. Τελικά καταφέραμε να προσαρμόσουμε τις τροπολογίες λαμβάνοντας υπόψη και τα συμπεράσματα αυτά. Σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Έτος για την ε, ενεργό γύρανση, είναι σημαντικό να επιμείνουμε στην αύξηση του προϋπολογισμού για τη χρηματοδότηση ε, του Ευρωπαϊκού Έτους. Και κυρία Πρόεδρε, αν εσείς δεν μπορείτε να υποστήριξετε την πρόταση, τουλάχιστον μην ε, την υπονομεύσετε. Ελπίζω η ψηφοφορία να είναι θετική για την τροπολογία αυτή. Σε ό,τι αφορά το συντονισμό το θέμα του συντονισμού είναι πολύ σημαντικό. Παρόλο που δεν συμφωνήσαμε σε όλες οι λεπτομέρειες, και θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες και στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. προσπαθώντας ε, να βρούμε ένα ρεαλιστικό τρόπο για να υλοποιήσουμε τις προτάσεις μας. Πάντως, όπως είπα και στην αρχή, γενικά συμφωνώ με τις προτάσεις της εισηγήτριας και την ευχαριστώ θερμά για, την, ε, για το έργο της. Ευχαριστώ κύριο Στέρκας. Κυρία Πρόεδρε, και οι σοσιαλιστές θα υποστηρίξουν τη γνωμοδότηση στα δύο θέματα και την γνωμοδότηση και της τροπολογίας. Ακούσαμε τις προτάσεις και συμφωνούμε μαζί σας ότι διανύουμε μια ιστορική στιγμή στην Ευρώπη και απαιτείται από εμά μια συνέπεια που είχαμε δείξει ούτως ή άλλως και δείχνουμε και είχαμε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση με το Συμβούλιο προσπαθώντας να συμφωνήσουμε ώστε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη για να αξιοποιήσουν καλύτερα τα κονδύλια που έχουν στη διάθεσή του και να αντιμετωπίσουν τι δυσκολίε, χρειαζόμαστε συνέπεια, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλισμό. Και ρεαλισμό σημαίνει να μείνουμε κοντά στο κείμενο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα ποσά και στη σκέψη τη, ώστε να καταλάβει και το Συμβούλιο ότι και η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια σε επαγγελματισμό και υπευθυνότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα στηρίξουμε τις τροπολογίες σας. Και εγώ θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την πρόταση. Χωρίς μικρόφωνο η πρόεδρος δεν ακούγεται. δεν σας είχα δώσει το λόγο λέει προφανώς. Κανένα πρόβλημα. θα μπορούσε πρώτα να μιλήσει η κυρία Χάρκιν κάλλιστα και εγώ μετά. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι οι προτάσεις της ΓΚΟΕ λαμβάνουν υπόψη μια διαφορετική πραγματικότητα, αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε στις πατρίδες μας. Μια κοινωνική κατάσταση με επιδείνωση με της φτώχειας, της ανεργίας και άρα ανάγκης για πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη στον κοινωνικό τομέα. Βέβαια, όντω, οι προτάσει μα δεν λαμβάνουν υπόψη την, οικονομική, την δημοσιονομική πραγματικότητα, την πραγματικότητα του προπολογισμού. Δυστυχώ αυτή η δημοσιονομική πραγματικότητα μα οδηγεί σε ένα αδιέξοδο, γιατί δεν λαμβάνει υπόψη την επιδείνωση των ανισοτήτων και την όξυση τη κοινωνική κατάσταση ε, που διαπιστώνουμε σε πολλέ χώρε, μεταξύ άλλων και στην Πορτογαλία. Γι' αυτού του λόγου, λοιπόν, εμεί ε, διεκδικούμε μια πολύ μεγαλύτερη προσοχή στα κοινωνικά ζητήματα. Βέβαια, αντιλαμβάνομαι τη θέση της εισηγήτριας που είπε ότι η πρότασή μας δεν είναι ρεαλιστική. Δεν είναι ρεαλιστική στο πλαίσιο του προϋπολογισμού μας, αλλά είναι ρεαλιστική γιατί λαμβάνει υπόψη την πραγματική κατάσταση, την κοινωνική κατάσταση που βιώνουμε σε πολλές χώρες και στη δική μου, την Πορτογαλία. Αυτή την διαφοροποίηση θα ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ. Θα είμαι λοιπόν πάντα σύντομη. Υποστηρίζουμε τα δύο ντοσιέ. Κάποιες μικρές παρατηρήσεις για τη γνωμοδότηση. Εγώ προτιμώ τον όρο κατάλληλος προϋπολογισμός και όχι αύξηση του προϋπολογισμού. Αλλά δεν συμφωνώ με την τροπολογία Χέλμερ που λέει ότι η κρίση έχει ήδη περάσει. Σχετικά τώρα με την τροπολογία 17 για τις αξιολογήσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Οι αξιολογήσεις αυτές λειτουργούν ήδη, οπότε δεν καταλαβαίνω την πρόταση δημιουργίας περαιτέρω τέτοιου είδους ενεργειών. Σχετικά τώρα με τον ίδιο τον προϋπολογισμό, εμείς θα συμφωνήσουμε με την αποκατάσταση του προς υπόμνηση και θα υποστηρίξουμε μόνο επίσης την αύξηση για την ενεργή τρίτη ηλικία. Καλώς, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις, θα περάσουμε τώρα πλέον στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή τις ψηφοφορίες. Ελπίζω να έχετε όλοι τις κάρτες σας. Συνεπώς μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε πρώτα την γνωμοδότηση. Για την γνωμοδότηση αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι υποστηρίζω τις τροπολογίες 5 και 6 του κυρίου Χέλμερ εφόσον θεωρηθούν προσθήκες Εφόσον επιθυμείτε λοιπόν να ακολουθήσετε τις προτάσεις της εισηγήτριάς σας, από ό,τι βλέπω συμφωνείτε, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Έχω επίσης την τροπολογία ένα χέλμερ, είμαι κατά. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεν γίνεται δεκτή. Στην παράγραφο 1 έχω την 2 του κυρίου Χέλμερη με πάντα κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 της κυρίας Χάρκινγκ είμαι υπέρ ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παράγραφος 2 τροπολογία 5 Χέλμερ υπέρ σαν προστίκη ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Καταπίπτει η 4, η 6 θα μπορούσε να γίνει δεκτή σαν προθήκη, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 7 και 9 καταπίπτουν, θέτω σε ψηφοφορία την 8, Σρέτερ και Τούρινεν που είναι συμβατή, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, Κοιτάξτε, ηλεκτρονικός έλεγχος λοιπόν. Θα ακολουθήσει ηλεκτρονικός έλεγχος να βεβαιωθούμε ότι δουλεύουν και τα μηχανήματα και ότι έχετε όλοι τις κάρτες σας. Θα ψηφίσετε υπέρ αλλά δεν έχετε την κάρτα σας. Καλώς λοιπόν ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας. Δύο σοσιαλιστές επιπλέον συμμετείχαν προηγουμένως. Λοιπόν, τώρα τελειώνει η ψηφοφορία. 17 υπέρ, 18 κατά, μία αποχή. Δεν γίνεται δεκτή. Με μία ψήφο διαφορά. Κύριε Ιούξ, αργήσατε, αλλά όχι ότι θα άλλαζε τίποτα. Μετά την παράγραφο 2, παράγραφο 10 της κυρία Φιγκουερέδο. Εγώ προτείνω αποχή, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Φτάνουμε τώρα στους συγκεκριμένους αριθμούς για μια στιγμή. Μετά την παράγραφο 2 μια προφορική τροπολογία της κυρίας Τούρινεν, την οποία γραπτά ενημερωθήκατε, είμαι υπέρ και είναι υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Στην παράγραφο 3 υπάρχει η τροπολογία 11, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 15 υπέρ 23 κατά είναι σαφές ότι δεν περνάει. Τροπολογία 12 των Πρασίνων. Ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 4 έχω την τροπολογία 13. Είμαι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά την παράγραφο 4 έχω την 14, ποιοι είναι υπέρ. Δεκτή. 15 είμαι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά α, δεκτή. Τροπολογία 16, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Στην παράγραφο 5 έχω την 17 Έλμερ, που είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 συνθετικό πνεύμα του Έλμερ, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 7. Έχω την 19 Χέλμερ. Είμαι κατά ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Την τροπολογία 20 είμαι κατά. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 20. Ψηφίσατε όλοι. Κύριε Ρέκνερ, ψηφίζετε κατά, δεν έχετε την κάρτα σας. Λοιπόν, 17-17 δεν γίνεται δεκτή. 21 του κυρίου Χέλμερ, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Μετά την παράγραφο 8 έχω την 22 του Ρίναν, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα για το σύνολο πλέον Άρχεται η ψηφοφορία, ψηφίσατε όλοι, κυρία Ρέγνερ ψηφίζει υπέρ, πέρας της ψηφοφορίας, 25, 35 ε, υπέρ μάλλον, κανείς κατά δύο αποχές, η γνωμοδότησή μας πλέον είναι έτοιμη. Περνάμε τώρα στο σημείο 5. Θα ψηφίσουμε αριθμούς τώρα πλέον. Euh, λοιπόν, θα περάσουμε τώρα, αν θέλετε, στο πιο περίπλοκο σημείο του προϋπολογισμού. Θα ξεκινήσουμε με την 6.617 και θα ψηφίσουμε πρώτα τους αριθμούς. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Ξαναρχίζουμε. Λοιπόν, 6.627 διορθώνει η πρόεδρος. Ποιοι είναι υπέρ των αριθμών. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεν γίνονται δεκτοί. Τα σχόλια καταπίπτουν. Ψηφίζουμε τώρα την 6.632 για τους αριθμούς, την αποκατάσταση δηλαδή του εγκειμένου της Επιτροπής. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 6.611 όροι, η καταπίπτη. Ψηφίζουμε τώρα την 6.612, τους αριθμούς του κυρίου όρη πάντα. και είναι υπέρ εγώ είμαι κατά. Ξαναρχίζω. Ποιοι είναι υπέρ της 6.612. Ποιοι είναι κατά. Ποιοι απέχουν. Δεν γίνεται δεκτή. 6.634. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεκτή, συγγνώμη λέει, πρόεδρος δεκτή. 6-6-35 ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Κατά. Δεκτή. 6 600... Α, θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για το 66-35. Ψηφίσατε όλοι, κυρία Ρέγνερ ψηφίζει υπέρ. 22 υπέρ 16 κατά ξεκάθαρα υιοθετηθήσα. Λοιπόν, η 13 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η 66-36 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66-37 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66-38 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66-14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66-59 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 66-39 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 66-74 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66-65 ποιοι είναι υπέρ κατά, αποχές, δεκτή, υπέρ. Για μια στιγμή. Την 66-63 μαζί με την προφορική τροπολογία που προβλέπει να προσθεθούν ορισμένα χρήματα. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τώρα οι τροπολογίες 66-21 και 66-40 είναι ταυτόσιμες αλλά έτσι και καταπίπτουν γιατί υπερψηφίσαμε την 63. Ψηφίζουμε λοιπόν τώρα την 66-22 η οποία έχει μόνο παρατηρήσεις. Ποιοι είναι υπέρ των παρατηρήσεων. Κατά αποχές δεκτές η τροπολογία 6603 Έρη και 6641 της εισηγήτριας είναι ταυτόσιμες, ψηφίζονται από κοινού ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Το ίδιο συμβαίνει και με την 6615 και την 6642 ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. Τρομολογία 6675 66-75 Φιγουερέδο, ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογίες 66-16 και 66-44 ταυτόσημες ποιοι είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτές 66-62 και 66-04 Α όχι δεν είναι ταυτόσημες. 62 πρώτα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 6604 καταπίπτει. Θέτω σε ψηφοφορία πλέον την τροπολογία τα σχόλια για το ΕΡΕΣ με την 6623. για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν των σχολείων, υπέρ κατά δεκτά. Τώρα 66-64, ποιοι είναι υπέρ κατά ποχές δεκτή. Φτάνουμε στην 66-06 με μία προσθήκη. είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα επαληθεύσουμε το 06. Έλεγχος για το 06. Ψηφίσατε όλοι. 21 υπέρ, 15 κατά, 2 αποχές. Δεκτή η τοπολογία. 6607 αποσύρθηκε φέτος σε ψηφοφορία την 6624 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Στην τροπολογία τώρα 66 ή 28 θα πρέπει να ψηφίσουμε μια θέση σε αποθεματικό. Ε, ο εισηγητής σας είναι κατά, ποιοι είναι υπέρ. Κατά Αποχές. Νομίζω ότι έγινε δεκτή. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά νομίζω ότι έγινε δεκτή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρα στις ψηφοφορίας. 20 υπέρ 15 κατά. Πράγματι λοιπόν γίνεται δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα το σχόλιο με μια προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ αυτής της προφορική τροπολογία κατά, υπέρ, ξανα, ξαναψηφίζουμε, κατά, αποχές, το σχόλιο συνεπώς δεν γίνεται δεκτό. Η τροπολογία 6029 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε τώρα τη συμβιβαστική τροπολογία α κεφαλαίο. Για τους αριθμούς πρώτα ποιοι είναι υπέρ των αριθμών δεκτή, τα σχόλια ποιοι είναι υπέρ των σχολείων, υπέρ κατά αποχές δεκτέ, δεκτά μάλλον. Τώρα η 66-30 καταπίπτει. Ερχόμαστε τώρα στη συμβιβαστική β για τους αριθμούς. Ποιοι είναι υπέρ κατά δεκτή. Για τα σχόλια υπέρ κατά αποχές δεκτά. 66.31 31 καταπίπτει, περνάμε τώρα στην 66-17. Είμαι υπέρ, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές 6673 66-73 καταπίπτει, 66-25 καταπίπτει επίσης. Αλλά αντίθετα θα πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια στο 66-25, ποιοι είναι υπέρ των σχολείων της κυρίας Τούρινεν. Κατά αποχές δεκτά τα σχόλια. Περνάμε τώρα στην 667 καταπίπτη, 6646 αποσύρθηκε, ψηφίζουμε την 6618 τσάμπα όρη. Είμαι υπέρ, είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66 τώρα 71. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 66 26 Τους αριθμούς, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτέ, τα σχόλια υπέρ, κατά, αποχές, δεκτά. Φτάνουμε τώρα Στην 66, 72, ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Η 66-69 καταπίπτει ως προς τους αριθμούς, αλλά πρέπει να ψηφίσουμε τα σχόλια. Λοιπόν, ποιοι είναι υπέρ των σχολείων της 69. Κατά αποχές δεκτά. Η 66-20 καταπίπτει, το ίδιο συμβαίνει και με την 66-48. Ψηφίζουμε τη 49 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66-60 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 61 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 66-50 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 6608 και 51 ταυτόσημες μαζί, ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές, 6670 για τους αριθμούς υπέρ κατά αποχές δεκ, απορρίπτονται, τα σχόλια καταπίπτουν πλέον. Η 6600 έχει καλυφθεί από τη συμβιβαστική α, η 601 ε, το ίδιο με τη συμβιβαστική Β, η 6609 και η 6653 Είπαμε ότι η 6601 επειδή ψηφίσαμε τη συμβιβαστική Β καταπίπτει. Ψηφίζουμε τη 09 και την 53 λοιπόν ποιοι είναι υπέρ κατά αποχές δεκτές. 6654 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 66-58 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 66-55 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 66-02 τους αριθμούς, ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτή και τα σχόλια με την προφορική τροπολογία που είπα για την ενσωμάτωση της πρότασης του κυρίου Μπουλό για το επιχειρηματικό πνεύμα και την καινοτομία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτά τα σχόλια. 66-66 καταπίπτει, 66-56 απεσύρθη, 66-57 ποιοι είναι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτά. 66-10 και 52 ταυτόσημε Στη θέτω από κοινού σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά αποχές δεκτές τελειώσαμε με τους αριθμούς αλλά όχι με την τελική ψήφο. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σας προτείνω να ψηφίζουμε en bloc τις επιστολές για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση 1, 2, 3, τέσσερις ε, περιπτώσεις Ολλανδικές δεν υπάρχει κάποιος κατά. Ψηφίζουμε en bloc αυτές, αυτά τα τέσσερα γράμματα υπέρ, κατά, δεκτά σχεδόν ομόφωνα με κάποιες όμως διαφοροποίησεις. Σας ευχαριστώ όλους και θα παραχωρήσω τώρα την Προεδρία στον πρώτο Αντιπρόεδρο, στην πρώτη Αντιπρόεδρο, την κυρία Λίνη. Η έκθεση του κυρίου Νταντέν είπαμε θα συζητηθεί ε, τον Οκτώβριο, 6 Οκτωβρίου αλλά θα συζητήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, δεν ε, θα υπάρξει ψηφοφορία είναι διότι οι τροπολογίες δεν ήταν ε, αγγλικά και πολλές ομάδες πρέπει να διασφαλίσουν ότι η ψηφοφορία θα γινόταν ορθώς. Οπότε ευχαριστώ τον κύριο Νταρντέν που έλαβε το θέμα αυτό υπόψη και δέχτηκε να υπάρξει μία αναβολή τις ψηφοφορίες. Θα ήθελα όμως να συζητήσουμε τις συμβιβαστικές τροπολογίες και όπως σας είπα έχει καθυστερήσει ή ε, ε, έχει αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι τις 6 Οκτωβρίου. Ο κύριος Νταρντέν. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα αναφερθώ στο timing και στις διαδικασίες και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή διότι πιστεύω ότι θα συμβάλλει εις ε, την ε, ποιότητα της εκθέσεως και αυτό είναι βασικό και υπήρχαν διάφορα θέματα και ιδίως η μετάφραση για να μπορέσει να ε, συζητηθεί ε, και να αναλυθούν οι διάφορες συμβιβαστικές. Θέλουμε όμως ε, το χρονοδιάγραμμα να είναι λογικό. Δηλαδή να είναι ένα χρονοδιάγραμμα το οποίο θα επιτρέψει να υιοθετήσουμε ελπίζω οι αρχές Οκτωβρίου ή στην Επιτροπή το σχέδιο αυτό εκθέσεως. Οπότε ακόμη και αν στην Ολομέλεια η, η ψηφοφορία γίνει τον Νοέμβριο δηλαδή μετά από την πρώτη σύμβαση για, στην Κρακοβία για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα που ε, θα γίνει τον Οκτώβριο. Ε, ελπίζω ότι εντωμεταξύ θα το έχουμε ε, τουλάχιστον υιοθετήσει σε επίπεδο επιτροπής. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία ε, γιατί πρέπει να δώσει ένα μήνυμα προς τα έξω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διότι επί της ουσίας νομίζω ότι στα πλαίσια της ε, ε, συνολικής καταστάσεως της οικονομικής κρίσεως την οποία βιώνουμε πρέπει να διακηρύξουμε μέσω της εκθέσεως αυτής ότι δεν μπορεί να πάει σε δεύτερη μοίρα το θέμα που μας απασχολεί και αυτοί οι βασικοί στόχοι ε, πρέπει να επιζητηθούν ε, εκ του παραλίλου και γι' αυτό είναι βασικό διάφορα θέματα τα οποία έχουν ε, εξεταστεί από την Επιτροπή αυτή σε συγκεκριμένες εκθέσεις να επαναληφθούν και να ανακεφαλαιωθούν στα πλαίσια αυτής της εκθέσεως για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά τρόπο ώστε να υπάρξει μία προστιθέμενη αξία μέσω αυτής της εκθέσεως. Μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα νομίζω ότι η έκθεση αυτή εξετάζει την περίοδο μέχρι το 2020 και γι' αυτό μπορεί να περιλάβει στόχους οι οποίοι ίσως ε, είναι λίγο πιο μακριά από αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί εις ε, τις ε, συγκεκριμένες εκθέσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι αν δεν κάνουμε επιπλέον βήματα προς τα εμπρός θα δεν θα είναι θετικό αυτό και για μας και για όλους τους παρατηρητές από πλευράς πρακτικής 396 τροπολογίες δηλαδή υπήρχαν πάρα πολλές τροπολογίες που είχαν υποβληθεί πράγμα που δείχνει τι ενδιαφέρον προκαλεί το θέμα αυτό έχουμε συντάξει συμβιβαστικές προτάσεις περίπου 45 δηλαδή κάποια πενινταριά συμβιβαστικών ισεών για 230 ε, τροπολογίες εκ οι οποίες αφήνουν δηλαδή ακόμη προσυζήτηση περίπου 130-140 αλλά μπορούμε έτσι να ε, συνοψίσουμε ορισμένες τροπολογίες και οι περισσότερες από αυτές τις συμβιβαστικές λύσεις είναι αντικείμενο με ευρεία συνένεση. Και εδώ Σκέφτομαι ιδίω τις ανάγκες να προωθήσουμε την εργασία των νέων, προστασία των ευαλώτων ομάδων όπως οι ηλικιωμένοι, οι πολλοί νέοι, διότι εδώ υπάρχει συνένεση όλων των οργανώσεων που ασχολούνται με τις ομάδες αυτές για την καταπολέμηση της φτώχειας, υπάρχει ο ρόλος της σημασίας στο θέμα της κατοικίας Νομίζω ότι όλα αυτά δεν θα ε, προβληματίσουν ε, διότι ήδη έχουν συζητηθεί με τους συντονιστές ε, στα θέματα αυτά και ελπίζω θα πάμε καλά. Υπάρχουν όμως και διάφορα ακαθόδη σημεία τα οποία είχαν τονιστεί όταν παρουσιάστηκαν οι τροπολογίες. Έχω όμως ότι τελικά θα, θα πιστεύω ότι θα μπορέσουμε τελικά να συμφωνήσουμε και ε, σχετικά με ε, ό,τι έχει καταλήξει σε μία συνένεση θα μπορέσουμε ε, να συμφωνήσουμε. Δηλαδή το ελάχιστο εισόδημα όπου υπάρχουν αντιγνωμίες και όπου έχω διατυπώσει μία ενδιάμεση πρόταση για διαβούλευση της Επιτροπής σχετικά με την ανάγκη μίας νομοθετικής Θα προσπαθήσουμε να ε, την προωθήσουμε. Υπάρχει το ε, το, το ε, νομοθετικό πλαίσιο της ε, καλύψεως ορισμένων ομάδων, ε, οριζόντιες συζητήσεις, επανερχόμαστε και η σχέση μεταξύ οικονομίας και φτώχειας ε, στα πλαίσια της οικονομικής διακυβέρνησης, όλα αυτά πρέπει να βελτιωθούν όσον αφορά τη σύνταξη, κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε λύσεις στα θέματα αυτά, αλλά πρέπει να σας πω ότι μέχρι στιγμής έχω την άποψη ότι οι συζητήσεις έχουν καταλήξει καταλήξει επικοδομητικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος ο οποίος θέλει να αναφερθεί σχετικά ε, σε αυτό το σημείο. Η κυρία Φιγκερέντο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Νταρντέν εκπώνησε με τους συνεργάτες του ένα αξιόλογο θετικό έργο προσπαθώντας να βρει έναν όσο πιο ευρύ ελάχιστο κοινό παρανομαστή γίνεται μεταξύ των διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και στο πλαίσιο αυτό αντιλαμβανόμαστε και την πρόταση αναβολής της ψηφοφορίας. Μάλιστα, πολλοί βουλευτές ε, συντάχθηκαν με αυτή τη θέση της αναβολής, γιατί υπήρχαν προβλήματα μετάφρασης ε, πολλών τροπολογιών και συμβαστικών λύσεων και είναι σημαντικό να περιμένουμε και να διαβάσουμε στις γλώσσες μας αυτές τις συμβαστικές προτάσεις ε, με ζητούμενο την συνένεση στη, στον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Φυσικά υπάρχει διάσταση απόψεων που οφείλεται όχι τόσο στην διάγνωση που κάνουμε και στην ανάλυση της επιδείνωσης της φτώχειας και της αόξυνσης των ανισοτήτων, η διαφορά απόψεων προκύπτει κυρίως από τις διαφωνίες που έχουμε ως προς τις αιτίες αυτής της επιδείνωσης της κατάστασης και της όξυσης της φτώχειας. Ε, εκείνη που υπάρχει διάσταση απόψεων, ως προς τα αίτια του κακού. Και είναι γνωστό άλλωστε αυτό. Υπάρχει αυτή η διχογνωμία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και θα φανεί και στην ψηφοφορία ορισμένων τροπολογιών. και στις διάφορες συμβαστικές λύσεις, που μερικές είναι πιο συνενετικές από άλλες. Πάντως, τα αίτια της φτώχειας δεν έχουν καταπολεμηθεί ακόμη. Εξακολουθούν να υπάρχουν και μάλιστα εντείνονται. Γι' αυτό οξύνεται και η φτώχεια, γι' αυτό επιδεινώνονται και οι ανισότητες. Αυτό είναι και το πρόβλημα των λεγόμενων σχεδίων λιτότητες. Η Πορτογαλία, η πατρίδα μου, έγινε θύμα αυτής της κατάστασης και μάλιστα όχι μόνο εξαρθρώνονται, τα υπολείμματα του υποτιθέμενου κράτους πρόνοιας, αλλά φτάνει σε ανησυχητικές και εξοργιστικές διαστάσεις ε, το φαινόμενο της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων. Και δυστυχώς η έκθεση αυτή δεν καταφέρει να δώσει μια λύση στην κατάσταση, γιατί η λύση θα προέλθει από άλλες πολιτικές που δυστυχώς δεν μεταρρυθμίζονται με τον τρόπο που χρειάζεται. Γι' αυτό και ναι, μεν η θέση μας είναι θετική και η εκτίμηση της ε, έκθεσης είναι θετική. Απ' την άλλη, ε, επικρίνουμε τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιμένουν σε αποφάσεις και καταστάσεις που επιδεινώνουν τη φτώχεια και τις κοινωνικές ενισότητες. Ευχαριστώ. Η κυρία Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας που πραγματικά συνεργάστηκε θαυμάσια με τους σκιώδεις εισηγητές. Αλλά πραγματικά λυπούμε ειλικρινά για την αναβολή της ψηφοφορίας παρά την επίγουσα κατάσταση. Ακριβώς λόγω του προβλήματος, του ατυχούς προβλήματος που είχαμε με τις καθυστερήσεις της μεταφράσεις. Νομίζω ότι Είναι μια στιγμή όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλείται να υπενθυμίσει το ρόλο του λίγο πριν την πρώτη συνδιάσκεψη που θα γίνει στις 16 Οκτωβρίου για τη συνένεση. Έπρεπε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα. Ενώ τώρα με την αναβολή θα περιμένουμε και η έκθεσή μας δεν θα υποβληθεί πριν αυτή τη διάσκεψη της συνένεσης. Δυστυχώς. Σε ό,τι αφορά την έκθεση. Δεν έχω ιδιαίτερε αντιρρήσεις. Νομίζω ότι το ζήτημα τη φτώχεια θα πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να αντιληφθούν πω απέναντι στην οικονομική κρίση και απέναντι στην κοινωνική κρίση έχουμε ένα καθήκον και μια ευθύνη να προστατεύσουμε του πιο ευάλωτους συμπολίτε μα και να μην του αποκλείσουμε από τι κοινωνίε μα. Δυστυχώς δεν ε, παρέχουμε τη δέουσα αρρωγή ε, στους πιο ευάλωτους πολίτες. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι απλώς να τους βοηθήσουμε, αλλά να τους ε, βοηθήσουμε να εξασφαλίσουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την ισότητα δικαιωμάτων ως προς τη στέγαση, ως προς την εργασία, ως προς την πρόσβαση στις κοινοφελείς υπηρεσίες. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε μια πραγματικά κοινωνική Ευρώπη. Και ελπίζω αυτή η έκθεση να είναι ε, το πρώτο ορόσημο αυτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παροτρύνει τα κρατημέλη να στραφούν προ αυτή την κατεύθυνση τη δημιουργία μια αναβαθμισμένη κοινωνική Ευρώπη. Θα ήθελα κι εγώ, και και συγγήτρια της, ε, το φιλελευθέρω τη Άλντε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή μα για το συνεργάσιμο πνεύμα που επέδειξε και τη διαλεκτικότητά του. Πολύ αξιόλογη έκθεση και είναι σημαντικό να συντονιστούμε για να τη δώσουμε ένα σωστό περιεχόμενο και Χαίρομαι για την προσπάθεια που γίνεται να βρεθούν συμβαστικέ λύσει. Όλοι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα των αστέγων, τη φτώχεια σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Συμφωνώ με την κυρία Ντελή ότι κρίμα που δεν α, ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι μεταφράσεις ώστε να ψηφίσουμε εμπρόθεσμα και να διαβάσουμε την έκθεση πριν αυτή την διάσκεψη. Αλλά παρόλα αυτά θα παραμείνει φτώχεια στο κοινωτικό πρόγραμμα για πολύ καιρό, γιατί έχουμε στις 16 την ε, δράση για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επίσης ε, θα έχουμε ε, την ψηφοφορία τον Οκτώβριο και δεν ξέρω σε ποια ολομέλεια του Νοεμβρίου θα μεταβιβαστεί αυτή η έκθεση. Οπότε θα μείνει το θέμα στο πρόγραμμα για πολύ περισσότερο καιρό με αυτή την αναβολή. Έχω και μερικά σχόλια που τα κάναμε και στην συνεδρίαση των συντονιστών. Διαφωνώ με την κυρία Φιγκερέδο ότι αφορά τα μέτρα λιτότητα. Εγώ δεν πιστεύω ότι τα μέτρα λιτότητας πρέπει να τα κρίνουμε επικριτικά ή με τέτοιο, με τέτοιο πνεύμα. Είναι μια πραγματικότητα, είναι μια αναγκαιότητα. Και χαίρομαι που στο συμβαστική πρόταση L διευκρινίσω ότι δεν είναι μόνο οι γυναίκες που φέρουν αυτή την ευθύνη της φροντίδας, αλλά και οι άντρες, ειδικά όταν μιλούμε για τους γονείς. Και το γυναίκες να το αντικαταστήσουμε από το άνθρωποι. Στο Νίνι δεν ξέρω αν θα το συμπεριλάβετε τελικά. Είπαμε ότι το 128 θα είναι προσθήκη στη συμβαστική λύση και ίσως τελικά συμφωνήσει και ο εισηγητής. Τώρα για την διανομή τροφίμων θα το εξετάσουμε πιο λεπτομεριακά, αλλά περιμένουμε την αγγλική μετάφραση. Ήταν πολύ δύσκολο για μας που έχουμε τα αγγλικά, παρόλο που είχαμε τις μεταφράσεις και πραγματικά με βοήθησε πολύ και το, με βοήθησε πολύ και η αλλά ακριβώς ε, επειδή το πρωτότυπο δεν είναι το αγγλικό, θα πρέπει να είμαστε πολύ σχολαστικοί, γιατί μερικές φορές και μία λέξη και ένα μικρό λάθος μπορεί να αλλάξει τελείως το νόημα, μία μικρή διαφορά. Στο πι μιλάτε για τη συγχρηματοδότηση. Και εκεί έχουμε κάποια μικροπροβλήματα. Και το αίτημα για την οδηγία πλαίσιο. Είναι σημαντικό... Διακόπτη πρόεδρος. Είναι σημαντικό να μην έχουμε έτοιμα για μια οδηγία πλαίσιο. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή λύση. Και αν αφαιρέσετε αυτό το σημείο, νομίζω ότι θα έχετε πολύ μεγαλύτερη υποστήριξη. Ό,τι αφορά την νομοθετική πρόταση για το ελάχιστο εισόδημα. Συμφωνώ με την πρόταση αυτή σε εθνικό επίπεδο. Το συζητήσαμε και επ' ευκαιρία της έκθεσης Φιγκερέντο Νομίζω μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αν έχουμε και πάλι έτοιμα για μια νομοθετική πρωτοβουλία για το ελάχιστο εισόδημα στην έκθεση αυτή, που κατά το λοιπόν είναι πολύ αξιόλογη, ελοχεύει ο κίνδυνος ε, πολλοί να την καταψηφίσουν εξαιτία αυτών των σημείων προτιμούμε να είναι συντριπτική η πλειοψηφία υπέρ της έκθεσης. Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι να την υποστηρίξουν για να τονίσουμε την προσπάθεια καταπολέμησης της φτώχειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να γίνει η έκθεσή σας πραγματικά ένα ορόσημο και ένα σημείο αναφοράς για να, να δει ο πολίτης τι θέλει να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να περιορίσει τη φτώχεια. Βέβαια έχουμε πολύ μακρύ δρόμο μπροστά μας, ώστε να ολοκληρωθούν οι μεταφράσει, ώστε να μπορέσουν όλο και περισσότεροι συνάδελφοι να λάβουν μέρος στις διαπραγματεύσει. Πάντως σα ευχαριστώ και πάλι για την προεργασία που κάνατε και για την ε, πολύ αγαστή συνεργασία που είχατε με τους κοιόδης συγκητέ. Ήταν πραγματικά εκπληκτικός ο τρόπος με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Κύριε Νταρντέν, αν δεν, δεν υπάρχουν άλλα σχόλια θα σας ξαναδώσω το λόγο να δευτερολογήσετε και να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο. Νομίζω ότι συντρέχουν πια οι προϋποθέσεις για να σημειώσουμε πρόοδο, ώστε πραγματικά αυτή η έκθεση να δώσει ένα ηχηρό μήνυμα Όντως, αν είχαμε προλάβει και ολοκληρώσει την ψηφοφορία πριν τις 17 Οκτωβρίου θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά τουλάχιστον στην Επιτροπή μας να εγκριθεί πριν ε, από τη 16 Οκτωβρίου, γιατί όντως είναι έτσι και έτσι χειρό το μήνυμα. Φυσικά θα εξαρτηθεί και από το περιεχόμενο της έκθεσης, αλλά νομίζω ότι διαφαίνεται μία επιθυμία να προτάξουμε αυτή τη, τον κοινό μας στόχο της καταπολέμησης της φτώχειας και της ανάγκης εξασφάλισης αξιοπρέπειας, όπως ακούσαμε από τις παρατηρήσεις. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, αν δεν κάνω λάθος, μέσα σε δύο εβδομάδες θα είναι έτοιμες οι μεταφράσεις. Οπότε θα ευθυγραμμίσουμε το αγγλικό με το γαλλικό κείμενο για να σεβαστούμε το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Και περνάμε στο επόμενο σημείο. Δεν είναι σίγουρο για το σε ποια ολομέλεια θα ψηφίσουμε, αλλά κατά πάσα πιθανότητα 6 Οκτωβρίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή. Επόμενο θέμα τη ημερησια διαταξη διάμεση αναθεώρηση Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2007. 2012 για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτριά μου, στην κυρία Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το δικαίωμα στην υγεία είναι θεμελιώδες δικαίωμα του Ευρωπαίου πολίτη που θα πρέπει να την χάνει εγγυήσεων νομικά δεσμευτικών σχετικά με την υγεία του, την ασφάλειά του και την αξιοπρέπειά του. Την διαπίστωση αυτή θα πρέπει να επιδιώξουμε να την κάνουμε πραγματικότητα όλοι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καιρός είναι να ασχοληθεί με το θέμα της ποιότητας της ζωής στην εργασία. Είμαι πεπισμένη ότι ζούμε μια βαθιά οικονομική κρίση και μια κοινωνική κρίση και γι' αυτό ακριβώς η πολιτική εξουσία θα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα να σταματήσει ο κόσμος να υποφέρει όταν δουλεύει. Όταν διαπιστώνει κανείς τον χώρο εργασίας σήμερα βλέπει ότι υπάρχει αύξηση των χρόνιων ασθενειών. Ψυχοσωματικές ασθένειες, ψυχοκοινωνικές όπως το στρες, ε, παρενόχληση, ε, συνεχείς κατηγορίες, παρατηρήσεις, περιθωριοποιήσεις, ε, μειώσεις της αξιοπρέπειας κτλ και υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι ζουν πραγματικά μοναχικά στη δουλειά τους και οι οποίοι δυστυχώς βλέπουν να χειροτερεύουν σε βάθος οι συνθήκες και οι σχέσεις τους στην εργασία και πολλές φορές οδηγούνται στην αυτοκτονία τους στον χώρο εργασίας τους και αυτό φυσικά επηρεάζει και τους συναδέλφους τους και όχι μόνο τις οικογένειές τους. Νομίζω λοιπόν ότι και ο καρκίνος που είναι βασικός λόγος νησιμότητας στην εργασία κάθε χρόνο στη Γαλλία, στην Ευρώπη συγγνώμη, 170.000 Ευρωπαίοι συνδέονται με θανάτους που οφείλονται στην απασχόλησή τους. Ξέρετε τι έγινε πρόσφατα με τα αγκουράκια και είδαμε ότι θα πρέπει να γίνουν τεράστιες προσπάθειες για να σωθούν οι ζωές όλων αυτών που εργάζονται στους κλάδους αυτούς. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Ασφάλεια 2007-2012 περιλαμβάνει καλούς στόχους. Έχει προχωρήσει σε κάποιους από αυτούς, αλλά δεν σας το κρύβω ότι δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένη από τη γενική πρόοδο. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις, υπάρχουν παραλήψεις, σαν παράδειγμα καμία επικοινωνία ανάμεσα στην πολιτική υγεία, στην εργασία και στις υπόλοιπες δημόσιες πολιτικές όπως η υγεία, η βιομηχανία, οι μεταφορές, η εκπαίδευση, η ενέργεια κτλ. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιοι είναι οι βιολογικοί και χημικοί κίνδυνοι στα πλαίσια της εφαρμογής των ουσιών REACH θα πρέπει να βάλουμε στόχους δεσμευτικούς, θα πρέπει να έχουμε σαν στόχο ένα επιθεωρητή ε, εργασίας για 10.000 εργαζομένους, όπως το συστήνει το Διεθνές ε, ε, Γραφείο, και πρέπει να υπάρξει καταμέτρηση του χρόνου εργασίας, του ατυπικού χρόνου, της νυχτερινής εργασίας, της διακεκομένης εργασίας, την οποία υφίστανται κυρίαρχα γυναίκες και παιδιά. Θα πρέπει να σώσουμε επίσης και τα κοινοτικά κεκτημένα στον τομέα της υγείας ε, και της ασφάλειας στην εργασία. Αυτό το κεκτημένο πρέπει να συνεχίσει να συμπληρούνται από φιλόδοξες οδηγίες σε συγκεκριμένα θέματα και σε συγκεκριμένες φάσεις. Θυμίζω επίσης ε, ότι ο προσωρινός χαρακτήρας της εργασίας είναι παράγον κινδύνου για τους εργαζομένους που έχουν χαμηλά εισοδήματα. Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων ιδιαίτερα στην υπεργολαβία που έχουν πολλά προβλήματα όπως μεταφορά βαριών, βαρέων βαρών, επίσης ψυχοσωματική κίνδυνη και αυτά τα κοινοτικά κεκτημένα τα οποία όπως είπα έχουμε θα πρέπει να συμπληρωθούν από οδηγίες φιλόδοξες ιδιαίτερα σε θέματα και σε συγκεκριμένους τομείς. είπαμε αυτό. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι οδηγίες αυτές έτσι ώστε να καταστεί πιο αποτελεσματικό και συνεκτικό το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Οι νομοθέτες δεν μπορούν από μόνοι τους να τα κάνουν όλα, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι κοινωνικοί εταίροι και οι ίδιοι εργαζόμενοι και αυτό θα πρέπει να αφορά όλους τους εργαζομένους ανεξαρτήτως του καθεστώτος στο οποίο εργάζονται. Τελειώνοντας θα ήθελα να πω ότι οι προσπάθειες για τη βελτίωση της υγείας στην εργασία προέρχεται από μια λογική από την οποία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Η προώθηση των πρακτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία είναι κάτι το ευεργετικό σε πολλούς τομείς. Ε, σε προσωπικό επίπεδο αλλά φυσικά επίσης και σε οικονομικό και σε κοινωνικό. Συνεπώς λοιπόν το σύνθημά μας είναι πάρα πολύ απλό, δεν υπάρχει τίποτα το μοιραίο όταν χειροτερεύει η υγεία και η ασφάλεια θα πρέπει ε, πριν από οτιδήποτε άλλο να υπάρχει πολιτική βούληση για τις εγγυήσεις προς τους εργαζομένους και είμαι βέβαιη ότι είστε διατεθειμένοι να δράσουμε από κοινού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την ε, συνάδελφο την Καρή Μαντελή για, μια, για αυτή την έκθεση που είναι πάρα πολύ καλή. Ε, κατά τη γνώμη μας ε, καλύπτει το μεγαλύτερο αριθμό των ζητημάτων. Είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να εργαστούμε και με βρίσκει σύμφωνη σχεδόν στα περισσότερα ζητήματα. Ε, θεωρώ υποχρέωσή μου να υπογραμμίσω ως εξαιρετικά θετικές ε, τις δύο προτάσεις για τις δύο νομοθετικές προτάσεις που κάνει. Η μία που αφορά τα ψυχικά νοσήματα και η δεύτερη που αφορά την προστασία των ε, όλων όσων εργάζονται με το καθεστώς της υπεργολαβίας. Ε, επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία να προστατεύονται οι εργαζόμενοι που καταγγέλουν παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας. Ε, τώρα, αισθάνομαι ότι θα είναι προς όφελος όλων αν έχουμε στο μυαλό μας επίσης ότι θα πρέπει να βοηθούμε τα κράτη-μέλη στο να εκπονούν καλύτερη νομοθεσία παρέχοντάς τους όλα τα απαραίτητα επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνεται η ανταλλαγή καλών πρακτικών να στηρίζονται οικονομικά όχι μόνο μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αλλά και από το 7ο ε, πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα ε, είναι εκεί που γίνεται αρκετή κουβέντα για πρωτοποριακές έρευνες και για πρακτικές που κατά τη γνώμη μου βοηθούν την καλύτερη εφαρμογή κανόνων για την ασφάλεια στην εργασία. Ε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαμε και αντίστοιχες εμπειρίες από το έκτο α, πρόγραμμα. Ένα άλλο θέμα πάρα πολύ σημαντικό είναι να συμμετέχουν, το υπογράμμισε η Καρίμα, ε, οι κοινωνικοί εταίροι και οι εργαζόμενοι στα συμβούλια που λαμβάνουν αποφάσεις σε σχέση με τα ζητήματα της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο των εργαζομένων. Ε, η συνεργασία και ο συντονισμός των διαφόρων ευρωπαϊκών οργανισμών και των Επιτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα θέματα του τομέα ασφάλειας στην εργασία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, νομίζω επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά των επιχειρήσεων ε, για σεβασμό συγκεκριμένων κανόνων ασφάλειας στην εργασία και η υποχρέωση αυτή μπορεί από από τη μια πλευρά να πρημοδοτείται με κίνητρα, αλλά από την άλλη μεριά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει και ποινή, όπως για παράδειγμα η επιβολή προστήμων. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη φροντίδα και μέρημνα στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων που, έχουν, που, που αφορούν άτομα με αναπηρία. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Όπως επίσης και με τους ανθρώπους που εργάζονται και ανήκουν στις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Ένα άλλο θέμα είναι ότι θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να προσαρμόζουμε τους κανόνες των δημοσίων συμβάσεων με τρόπο τέτοιο ώστε εάν είναι δυνατόν να πρημοδοτούνται εταιρείε που σέβονται και προωθούν τους κανόνες ασφάλειας και στηρίζουν τους εργαζόμενους σε θέματα υγείας. Ασφαλώς με ε, αποδείξεις. Ε, υπάρχουν πέρα από τους εργαζόμενους στα παραδοσιακά, να, το πω έτσι, επαγγέλματα, ε, υπάρχουν οι εργαζόμενοι στα επαγγέλματα και στις επιχειρήσεις που έχουν σχέση με την πρόοδο της τεχνολογίας. Παράδειγμα η νανοτεχνολογία ή παράδειγμα οι επιχειρήσεις που πια χειρίζονται ε, νέα χημικά, νέα βιολογικά προϊόντα. Αυτό είναι κάτι καινούριο που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ε, έχοντας στο μυαλό μας όχι μόνο το σήμερα, αλλά και το αύριο και το μέλλον. Ε, νομίζω ότι το να πω οτιδήποτε περισσότερο ε, θα κρατήσω το χρόνο σας χωρίς να προσθέσω κάτι περισσότερο στην πολύ καλή έκθεση που κατέθεσε η Καρή Μαντελή. Ε, κλείνοντας, θα κινηθώ σε αυτές τις γραμμές που περιέγραψα προκειμένου να καταθέσω τροπολογίες ε, βελτιωτικές και προωθητικές ακόμη περισσότερο έχοντας στο μυαλό μου πάντα την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων που εξασφαλίζουν την αξιοπρέπειά τους. Ε, ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και προσδοκώ μια εξαιρετική συνεργασία με την Καρίμα και όλους τους σκιώδες. Uh, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εκθερετική έκθεσή της που είναι ισοσκελισμένη και αρκετά πλήρης και παρόλα αυτά λόγω του αριθμού των σελίδων ε, πιστεύω ότι μπορούμε κάτι να προσθέσουμε σε αυτήν διότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιτροπών και θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι η κυρία Καρίμ Νταλή αναφέρεται ιδιαίτερο στην υπεργολαβία όπου έχουμε πολλά προβλήματα διότι η υπεργολαβία δεν πάει σε ε, μία υπεργολάβο επιχείρηση αλλά μετακυλάται ε, και σε άλλες οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να ελέγξουμε. Επίσης υπάρχουν οι διαφορετικές αντιμετωπίσεις στα διάφορα κράτη και είναι κάτι που πρέπει να ε, εξεταστεί σε αυτή την έκθεση και γι' αυτό θεωρώ ότι η συγκέντρωση των στοιχείων είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πρέπει να ασχοληθούμε με τις βέλτιστες πρακτικές και να είμαστε συνεκτικοί μεταξύ αυτής της πολιτικής και άλλων σχετικών θεμάτων. Δηλαδή κάπως θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρος σε αυτό το θέμα. Θεωρώ πολύ καλή και την ε, θέληση να ενισχύσουμε την επιθεώρηση εργασίας, τις υπηρεσίες επιθεωρήσεως εργασίας, γιατί μπορούμε να έχουμε θαυμάσια νομοθεσία, αλλά αν δεν υπάρχει μετά ε, έλεγχος και δεν υπάρχουν κυρώσεις, δεν μας ωφελεί να έχουμε την καλύτερη δυνατόν νομοθεσία. Επίσης αναφερθήκαμε στους κινδύνους για τις νέες τεχνολογίες και ιδίω τις νανοτεχνολογίες και πιστεύω ότι και στο σημείο αυτό πρέπει να μελετήσουμε πολύ περισσότερο διότι πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι τεχνολογίες του μέλλοντος με, όλους, τα θέματα τα οποία ε, συμπεριλαμβάνουν. Επίσης όσον αφορά το χώρο εργασίας όπως είπε και η συγγήτρια, υπάρχουν πολλά παραδείγματα για τη σημασία του θέματος αυτού με όλες τις αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις, τις αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία και για την οικογενειακή ζωή. Σχετικά με το σημείο 9 όμως, πιστεύω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε διότι θεωρώ ότι δεν είναι πολύ σαφές και πέραν αυτού θα ήθελα να σας πω ότι οι στατιστικές έχουν αποδείξει ότι σε πολλά σημεία υπάρχουν ατυχήματα, δηλαδή δεν είναι μόνο τα ατυχήματα στο χώρο συνεργασία αλλά και στο, ε, ε, οδό προς ή από την εργασία και θα πρέπει να ενισχύσουμε και την οδική ασφάλεια διότι σύμφωνα με τις διεθνείς στατιστικές βλέπουμε ότι και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ε, προσβλέπω στην συνεργασία και ε, πιστεύω ότι με τις προτάσεις θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και ε, ε, περιμένω με ανυπομονησία τις τροπολογίες. Ευχαριστώ ο κύριος Κοφεράτη και μετά ο κύριος Άσου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο ε, για το ενδιαφέρον και τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποίησε για να παρουσιάσει την πρότασή της και ε, ε, δίνω ιδιαίτερη σημασία εις ε, τη διάθεσή της να τα συζητήσει. Θα ήθελα να τονίσω ιδίω δύο θέματα, ιδίω την υπεργολαβία, διότι το θέμα αυτό έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ τελευταία και έχει οξυνθεί με την κρίση γιατί υπάρχουν πολλά συστήματα παραγωγής που χρησιμοποιούνται για να αντιμετωπιστεί ε, το κόστος ε, ε, διότι υπήρξαν δυσκολίες στην αγορά και πολλές φορές αψήφιστα χρησιμοποιεί κανείς την υπεργολαβία. Μεταξύ λοιπόν των θεμάτων των οποίων μπορεί κανείς να προωθήσει για να καλύψει τους εργαζομένους που εργάζονται σε αυτή στη μακριά αλυσίδα εκχωρήσεως των ευθυνών είναι να δώσουν δώσουμε τη νομική δυνατότητα στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων ή στους, ε, στις συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις των εργαζομένων να είναι καλά ενημερωμένοι σχετικά με τον τελικό στόχο της δραστηριότητας και να γνωρίζουν γιατί υπάρχει κάποια υπεργολαβία. Επιπλέον στη συνέχεια καταλήγει κανείς εις ε, τον καθορισμό ενός ε, συγκεκριμένου αγαθού διότι ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε κάθε κίνδυνο στα θέματα υπεργολαβίας. Επίσης πολλές φορές θεωρούμε ότι η πρόληψη αναφέρεται ιδίω στα άτομα και τους κινδύνους που αναλαμβάνουν τα άτομα αυτά. Αλλά όταν ένα προϊόν ή ένας τρόπος παραγωγής ε, υπάρχει ήδη, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε την ασφάλεια από την πρώτη στιγμή που ο σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα εκ προημίου και όχι εκ των υστέρων διότι οι νέες παραγωγές ε, σχετικά με τον τρόπο παραγωγής σημαίνουν ότι μπορούν να ληφθούν, διατακ, ε, ληφθούν μέτρα για να μειωθούν οι κίνδυνοι και πρέπει να ληφθούν υπόψη από την αρχή κατά τρόπον ώστε να ενθαρρύνουμε από την αρχή την ε, έρευνα σχετικά με την ασφάλεια. Συνεπώς αυτή η υπόθεση νομοθετική η οποία έγινε μπορεί να υπάρξει μια συγκεκριμένη αναφορά στις δραστηριότητες τις προγραμματικές και τις ερευνητικές τις οποίες έχουμε μπροστά μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Χέρς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, προσωπώ τον ισχυρό δισηγητή κύριο Κρόιτσμαν που δυστυχώς δεν παρίσταται. Καταρχήν όμως ευχαριστεί για την καλή συνεργασία, την καλή έκθεση διότι η ασφάλεια στο χώρο της εργασίας και η υγεία είναι πολύ σημαντικές για μας και γι' αυτό χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που γίνονται στον τομέα αυτό πρέπει να κινηθούμε στα πλαίσια των ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων και να τονίσουμε την επικουρικότητα. Δεν χρειάζεται μόνο νομοθετικό μέσο, διότι έχουμε δυνατότητα να επέμβουμε και με άλλους τρόπους, μέχρι στιγμής έχουμε πολλά επιτύχει όπως άλλωστε αναγνωρίζει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, βλέπουμε όμως ότι επανερχόμαστε στα εργατικά ατυχήματα και βλέπουμε ότι πολλά από αυτά οφείλονται εις την επιδεινόμενη ε, οικονομική κατάσταση. Ε, δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε κάτι τέτοιες σκέψεις, αλλά θέλουμε να υπάρχει συνοχή και κοινή προσπάθεια. Επιπλέον, το δικαίωμα για κοινή υγεία και ασφάλεια είναι ε, ενιαίο και διεθνές. Δεν ε, χρειάζονται μόνο ο νομοθετήματα που θα πέσουν στο κενό αλλά θα πρέπει ε, να εξηγήσουμε σε αυτούς οι οποίοι περνούν δύσκολες ε, ε, φάσεις ότι η προστασία της υγείας και η ασφάλεια της εργασίας συνεπιφέρουν και προστιθέμενη αξία. Διαφορετικά δεν θα τις αποδεχθούν και θα χάσουμε την ευκαιρία. Σχετικά με τις οριακές τιμές πρέπει να δούμε τι είναι ε, δυνατό τόνο και εφικτό ουσιαστικά διότι δεν μπορούν να υπάρξουν απλώς βελτιώσεις στη συνέχεια και τέλος δεν πρέπει να θεωρήσουμε απλώς ότι είναι ένας τομέας που γίνεται όλο και πιο σημαντικός αλλά πρέπει να αντιληφθούμε πώς και να κοιτάξουμε πώς θα λύσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται και να μην ε, λάβουμε στα γρήγορα αποφάσεις. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα να ερευνήσει σωστά το θέμα και μετά να προτείνει μέτρα. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτή είναι μια καλή βάση για περαιτέρω συζήτηση και θα εμπλακούμε προσπαθώντας να συνεργαστούμε και με τις άλλες πολιτικές ομάδες και χαιρετίζουμε τη συνεργασία αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους στόχους της έκθεσης αυτής που είναι πάρα πολύ σημαντική υγεία και ασφάλεια στην εργασία. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία θα πρέπει να τεθούν επιπλέον. Έχουν γίνει πολλές προτάσεις μέχρι τώρα για νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερη σημασία είναι να δούμε την εφαρμογή των υπαρχουσών ισχυρουσών οδηγιών και όχι να προτείνουμε νέε. Νομίζω επίσης ότι η σωστή διαχείριση των θεμάτων ασφαλείας και υγείας είναι πιο σημαντική από ε, περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, οι συγκεκριμένες υπάρχουσες οδηγίες να μπορούν να εφαρμοστούν σωστά. Είμαι λοιπόν αρκετά απογοητευμένοι από το θέμα αυτό, διότι δεν βρίσκω το λόγο να υπάρχουν νέες ε, ρυθμίσεις. Και δεν υπάρχει αναφορά στο ότι επίσης ε, οι ίδιοι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι επίσης για τα θέματα της ασφάλειας. Είναι, θα έλεγα, έχουν τον πιο σημαντικό ρόλο. Ε, σε ποιο βαθμό σέβονται τους κανόνες κτλ. Νομίζω ότι όλα αυτά θα πρέπει επίσης να αναφερθούν εδώ. και επίσης ε, χρησιμοποιεί κάποιες γενικές κατηγορίες όπως ε, η τηλεεργασία, οι υπεργολαβίες. Έχουμε διαφορετικές πολιτιστικές καταβολές και δεν μπορεί να πει κανείς ότι όλες οι, όλες οι δραστηριότητες στον τομέα της τελεεργασίας είναι κακές. Στις περισσότερες επιχειρήσεις στον τομέα αυτό το κλίμα, το περιβάλλον εργασίας είναι ίσως καλύτερο από άλλες μεγαλύτερες ε, επιχειρήσεις. Εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι καλή είναι η δουλειά την οποία έκανε η συγχύτρια και θα ήθελα να συνεργαστούμε μαζί της καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ, ο κύριος Αγαπητοί συνάδελφοι, Θεωρώ ότι η έκθεση της ε, συναδέλφου είναι μια θαυμάσια βάση και θέλω να τονίσω ότι ο συσχετισμός μεταξύ των μακρών ορών εργασίας και ανεπαρκή χρόνου ανάπευσης τονίζεται ικανοποιητικά στην έκθεση αυτή και γι' αυτό πιστεύω ότι ε, πρέπει να συμφωνήσω με τον κύριο Κρόιτσμαν ότι αν δεν υπάρχει επαρκής χρόνος αναπαύσεως για τους εργαζομένους οι οποίοι καταπονούνται πνευματικά ε, και σωματικά δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε. Ο χρόνος αναπαύσεως δεν είναι ε, ε, ένα δώρο, είναι αναγνώριση μιας ανάγκης και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι στην έκθεση ίσως θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την αξιολόγηση μιας εξελίξεως στις τελευταίας δεκαετίας στην Ευρώπη, δηλαδή βλέπουμε ε, μία μείωση ε, των μυϊκών ε, παθήσεων αλλά μία έκρηξη των ψυχολογικών και ψυχοσωματικών ασθενειών και πιστεύω ότι αυτή η διαπίστωση μπορεί να τονιστεί περισσότερο οπότε εγώ θα προβώ σε ορισμένες απολογίες επί του θέματος αυτού. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Περιμέναμε μια πολύ καλή έκθεση από τον συνάδελφο και δεν μας απογοήτευσε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δύο θέματα. Και να κάνω κάποιες διευκρινήσεις. Αναφέρθηκαν οι ευθύνες ε, των εργοδοτών. Φυσικά και ευθύνονται να, ε, να εφαρμόζουν σωστές πρακτικές υγείας και προστασίας. Το θέμα όμως είναι υπάρχει και γνώση και ποιες είναι οι προσδοκίες και των εργαζομένων σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Έχουμε πολλές νομοθετικές προτάσεις και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε εθνικό με επιπτώσεις ε, στην διαπαιδαγώγηση, στην παιδεία και στο σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στην προετοιμασία για τη δουλειά, ώστε ε, οι εργαζόμενοι να ξέρουν τι να περιμένουν, να ξέρουν ποιες θα είναι οι προσδοκίες τους. Μερικές φορές, ε, ειδικά οι νέοι, δεν γνωρίζουν καν ποιε θα πρέπει να είναι οι καλές πρακτικές στο χώρο, στο χώρο εργασίας. Οπότε τι να περιμένουν και πώς να κρίνουν αν γίνονται σεβαστές αυτές αφού δεν τις γνωρίζουν. Και το θέμα της γνώσης εκ μέρου των εργαζομένων είναι σημαντικό λοιπόν. Στο σημερινό εργασιακό κόσμο, ε, ο κόσμος αλλάζει πολύ πιο συχνά δουλειέ, είτε λόγω προσωπική επιλογή, είτε λόγω των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Και υπάρχει όλο και μεγαλύτερη πίεση ε, και στην, ε, στο χώρο εργασίας και στην όλη διαπαιδαγώγηση που θα πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Και όσοι έχουν ε, βραχυπρόθεσμες συμβάσεις και δουλεύουν ε, ε, λίγες ώρες, οι εργαζόμενοι που τους θέλουν γραφεία νεύρες εργασίες, αυτοί θεωρούνται ως εργαζόμενοι μερικές φορές δεύτερης κατηγορίας. Και υφίστανται καταστάσεις πολύ δύσκολες, καλούνται να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις. Για παράδειγμα, σε ένα ξενοδοχείο. Η μόνη δουλειά που μπορούσε να βρει κάποιο από γραφείο ανέβρε εργασία ήταν να καθαρίζει ε, του σε ένα μεγάλο ξενοδοχείο χωρί καν εξοπλισμό προστασία, χωρί καν γάντια, χωρί να έχει κάποια γνώση για τα τοξικά υλικά και διάφορα μέσα καθαρισμού που χρησιμοποιούσε. Θα πρέπει λοιπόν άσχετα με το χρόνο της ε, διάρκεια της σύμβαση και άσχετα από το αν ο εργαζόμενο προέρχεται από γραφείο, θα πρέπει να εξασφαλίζονται ίσε συνθήκες και υπάρχει θέμα διαχείριση. Μιλήσαμε και για το στρε στο χώρο εργασία. Πολλές επιχειρήσεις δεν ε, εφαρμόζουν πολιτική αντιμετώπιση ε, του στρες, του άγχου στην αγορά εργασία, ε, το να το εντοπίζουν, να το αναγνωρίζουν, να το διαχειρίζονται, ώστε να ελαχιστοποιούν το στρες, το άγχο τουλάχιστον στον χώρο τη εργασία. Γιατί φυσικά δεν μπορούμε να ελέγξουμε τη ζωή των εργαζομένων εκτό του χώρου εργασία. Και η διαχείριση και η κατάρτιση για τη διαχείριση του στρες είναι πολύ σημαντικό θέμα. Σε ό,τι αφορά την εργασιακή θεραπεία. Αυτή, ε, αυτό είναι πραγματικά ένα επάγγελμα των εργασιοθεραπευτών ε, που έχει τρομερές ελλείψεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, ε, συνήθως οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να καλύπτουν τα έξοδα της κατάρτισής τους. Δεν υπάρχει πρόβλεψη στο σύστημα υγείας για την κατάρτισή τους. Θα πρέπει λοιπόν να ενθαρρύνουμε όλο και περισσότερους ε, να ασχολούνται με θέματα υγείας στο χώρο εργασίας, γιατί πραγματικά αυτός ο τομέας ε, είναι αναπτυσσόμενος και νομίζω ότι όσο ε, γυράσκει το εργατικό δυναμικό θα χρειαστούν όλο και περισσότεροι επαγγελματίες στην υγεία της, στο χώρο της εργασίας. Κυρία Ντελή, αυτά που λέτε στην έκθεσή σα και για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πολύ σημαντικά. Εγώ ανέκαθεν πίστευα ότι εμεί ω Επιτροπή θα πρέπει περισσότερο να ασχολούθουμε με την εφαρμογή τη νομοθεσία στην υγεία και την ασφάλεια στην εργασία. Η Επιτροπή εσωτερική αγορά ασχολείται περισσότερο με το θέμα αυτό στη δική της, στο δικό του πλαίσιο αρμοδιοτήτων. Αλλά και εμεί έχουμε κάποιο λόγο να πούμε. Γιατί Είχαμε και διαδικασία συναπόφασης, οπότε συνομοθετούμε για πολλά θέματα, αλλά μερικέ φορές ε, δεν παρακολουθούμε μετά την ε, Παρασκευή της νομοθεσία, δεν παρακολουθούμε την εφαρμογή της. Θα πρέπει να δούμε, εφαρμόζονται όντω οι διατάξεις που εγκρίνουμε. Τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Η κυρία Εσάια είπε ότι πρώτα θα πρέπει να διαπιστώσουμε κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η υπάρχουσα νομοθεσία και μετά να προτείνουμε νέε νομοθετικέ προτάσει. Πρώτα να κάνουμε ένα απολογισμό τη εφαρμογή τη ισχύουσα νομοθεσία. Ίσως εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθεί και η Επιτροπή μας. Να παρακολουθούμε λοιπόν πώς δρομολογείται και πώς εφαρμόζεται μια νομοθετική πρόταση από την φάση της σύλληψης μέχρι τη φάση της εφαρμογής. Μιλήσατε σωστά για την υπεργολαβία, ιδιαίτερα την υπεργολαβία στον πυρηνικό τομέα. Και νομίζω ότι όντως είναι ένα θέμα που θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, να το επισημάνουμε. Μιλήσατε για το στρες, το άγχος και τα ψυχοκοινωνικά συμπτώματα. Για να δούμε στην πράξη τι μορφή θα μπορούσε να έχει μια τέτοια πρόταση. Υπάρχει και μια οδηγία για τις ε, μειοσκελετικές ε, διαταραχές, ε, αλλά νομίζω ότι αν προσθέσουμε σε αυτή την οδηγία το άγχος, κάπως θα την κατακαιρματίσουμε. Δεν νομίζω ότι θα είναι σωστή η αντιμετώπιση. Υπάρχουν πραγματικά ψυχοκοινωνικά προβλήματα αλλά αν τα συνδέσουμε με την οδηγία για τα μυοσκελετικά προβλήματα, θα δημιουργήσουμε ένα αμάλγαμα που δεν θα είναι αποτελεσματικό. Καλύτερα να διαχωρίσουμε τα δύο θέματα και αυτό να μην το θεωρήσουμε ως άλοθη για να αδιαφορήσουμε στο μέλλον για τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα προτιμώ η οδηγία για τη μειοσκελετικά προβλήματα να διαχωριστεί πλήρω από το μελλοντικό μα έργο ε, για το στρες, το άγχος στο χώρο εργασία ή τα κοινωνικοψυχολογικά προβλήματα στο χώρο εργασία. Κύριε Ντελή, φαντάζομαι ότι δεν θα, συμφωνώ, δεν θα συμφωνήσω μαζί σα ε, στην παράγραφο για την οδηγία που αφορά το χρόνο εργασία, ε, το ωράριο, αλλά φαντάζομαι ότι θα γίνουν αρκετά έντονη συζητήση για το θέμα αυτό στο μέλλον. Σας ευχαριστώ κύριε Ντέλη και έχετε το λόγο για τη δευτερολογία. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Διαπιστώνω ότι αυτό το θέμα παθιάζει πάρα πολλούς συναδέλφους, όχι μόνο εμένα, και χαίρομαι γιατί διαφαίνεται πολύ επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μας, χάρη σε αυτό το ενδιαφέρον. Πολλοί είπατε, τι περιμένουμε για να γίνουμε πιο αυστηροί, να είμαστε πιο απαιτητικοί απέναντι στις ε, εταιρείε και τις επιχειρήσεις αυτές που δεν τηρούν και δεν σέβονται τις διατάξεις υγείας και ασφάλειας για τους εργαζομένους τους. Αν θεωρείτε ότι δεν ήμουν αρκετά αυστηρή, παρακαλώ καταθέστε τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως να σα υπενθυμίσω ότι η βελτίωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας στην εργασία θα πρέπει να αποτελέσουν την προτεραιότητα ε, τη ευρωπαϊκή πολιτική. Βέβαια λένε μερικοί ότι έχουμε ισχύουσα νομοθεσία, γιατί να ζητήσουμε περισσότερα. Ζητάμε περισσότερα γιατί σήμερα στην οργάνωση της εργασίας υπάρχει μια αλλαγή. Διαπιστώνουμε μια αλλαγή, πολλά πράγματα έχουν τραποποιηθεί και γι' αυτό ζητούμε νέα νομοθεσία. Όχι για να επιβαρύνουμε την ισχύουσα νομοθεσία, και το νομοθετικό μηχανισμό, αλλά ακριβώς επειδή θέλουμε να βελτιώσουμε την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, θα θέλουμε αυτή την πρόκληση να την ε, αναγάγουμε σε σημαντική προτεραιότητα. Δεν θα σας υπενθυμίσω τα στοιχεία που σας έδωσα, αλλά δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε ε, σε αυτή την κατάσταση. Να ζητήσουμε πραγματικά ε, κέριους νομοθετικούς άξονες, γιατί το θέμα είναι επίγον λόγω της μεταβαλλόμενης κατάστασης και λόγω της οικονομικής αλλά και της κοινωνικής κρίσης. Έχουμε όλο και περισσότερη χρήση της μερικής απασχόλησης, έχουμε όλο και νέα προϊόντα στην αγορά. Μιλήσατε για τα πυρηνικά και θα ήθελα να επιμείνω στο γεγονός ότι το θέμα της υπεργολαβίας και ιδιαίτερα της αλλεπάλληλης υπεργολαβίας, γιατί σήμερα δεν έχουμε, ε, φτάνουμε με την υπεργολαβία σε 8 ο το επιπεδο και δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεργολαβία. Και οι εργαζόμενοι επίσης ε, τα έχουν χαμένα, γιατί αλλάζουν συνέχεια οι υπεργολάβοι. Γι' αυτό και θέλουμε να διατρανώσουμε αυτή την επιθυμία, να γίνει αυτή η νομοθετική πρόταση και το αίτημα σαφές ότι είναι και η ώρα να αναλάβουμε δράση. Σας ευχαριστώ. Ψάχνω εδώ το χρονοδιάγραμμα. Στις 16 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι λίγη προθεσμία για τις προθεσμίες. Θα συζητήσουμε τις τροπολογίες 6 και 7 Οκτωβρίου στην Επιτροπή. 7 Νοεμβρίου συμβαστικές λύσεις και στις 23 Νοεμβρίου θα εγκρίνουμε την έκθεση, θα ψηφίσουμε μάλλον την έκθεση στην Επιτροπή μας. Και προχωράμε στην επόμενη έκθεση που αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2005-36 σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Κάμπρνοχ. Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych krátce uvedl. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στις τροπολογίες οι οποίες έχουν υποβληθεί στην έκθεσή μου. Καταρχάς να ξεκινήσω ευχαριστώντας όσους έκαναν και κατέθεσαν τροπολογίες. 91 κατετέθησαν στην αρχή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον ε, για όλες και σε όλες τις πολιτικές ομάδες. Αυτό έχει σχέση με το ποσοστό ανεργίας, η οποία δεν είναι κυκλικό φαινόμενο, αλλά είναι κάτι το οποίο υπόκειται στην οικονομική συγκυρία. Να υπογραμμίσω επίσης ότι προετοιμάζουμε μία γνωμοδότηση προς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή που είναι η ίνκο στη συγκεκριμένη περίπτωση. συγκέντρωσα την προσοχή μου στα θέματα τα οποία μας αφορούν. Δεν μπορώ να κάνω δεκτό τροπολογίες που ασχολούνται με άλλα θέματα όπως ε, η ποιότητα της εργασίας, οι πράσινες θέσεις εργασίας, η διαβίου κατάρτιση. Είμαι υποχρεωμένος να συγκεντρώνω την προσοχή μου στον πυρήνα, αν θέλετε, της έκθεσής μου. Δέχομαι τις περισσότερες από τις τροπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί ε, και θα ε, τα συζητήσω αναλυτικότερα τα θέματα αυτά στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, ε, στις 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι στις 3 η ώρα με τους συναδέλφους και τους σκιώδεις εισηγητές. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλές τροπολογίες που εμπλουτίζουν την έκθεσή μου. Λίγες είναι αυτές τις οποίες δεν μπορώ να αποδεχτώ και δεν μπορώ να δεχθώ επίσης και τις τροπολογίες οι οποίες ε, ζητούν να υπάρξει περαιτέρω ε, νομοθετικές ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι δεν είναι κάτι τέτοιο απαραίτητο. για την 15 που αφορά την εξοχρονισμό των υπαρχουσών οδηγιών δεν υπάρχει πρόβλημα, η 20 που αφορά τη μείωση της γραφειοκρατίας, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία βελτιώνουν τη διαφάνεια, την πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Υπάρχουν επίσης και οι τροπολογίες 22 με 28 που στην ουσία αναφέρονται στη μείωση ενός αριθμού επαγγελμάτων, ρυθμίσεων μάλλον γύρω από συγκεκριμένα επαγγέλματα, ελεύθερα ή μη ελεύθερα. Υπάρχει επίσης η 54 και 58 που αφορά την κατάσταση συγκεκριμένων των οποίων έχει αφαιρεθεί η άδεια άσκησης επαγγέλματος και επίσης υπάρχουν γύρω στο 60 κάποιες τροπολογίες που αφορούν γλωσσικές γνώσεις. Υπάρχει επίσης μια δεύτερη ομάδα τροπολογιών ε, τις οποίες δεν πολύ καταλαβαίνω πολύ καλά θα είμαι ειλικρινής. Θέλω περισσότερες πληροφορίες όπως ε, γύρω από την 2. Πράγματι η Ευρώπη έχει ανάγκη ε, την κινητικότητα όλων των εργαζομένων και όχι μόνο των υψηλά εκπαιδευμένων και εξειδικευμένων. Δεν καταλαβαίνω επίσης τι ακριβώς θέλει η 32, πάντα στο θέμα της ε, κινητικότητας των εργαζομένων, όπως επίσης και της σύγκλησης των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει μια φυσική μορφή συντονισμού η οποία να βασίζεται στις υπάρχουσες πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι κάποια τεχνητή νομοθετική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βελτιώσει με οποιοδήποτε τρόπο τα πράγματα. Και θα συμφωνήσω με την τροπολογία Ουγγουρεάνου την 33 που ζητάει καλύτερο συντονισμό. Ε, πληροφορίες περισσότερες θέλω για την 35 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών ικανοτήτων και πτυχίων κτλ. Δεν την καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω και την έξι για την εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα ήθελα να θυμίσω ότι σε μια διαφορετική έκθεση είχαμε μιλήσει για το θέμα του συντονισμού των ε, συστημάτων αυτών και δεν μπορώ να δεχθώ την βασική αρχή ε, ε, της, που λέει ότι η ίδια, ίση αμοιβή, η ίδια αμοιβή για την ίδια εργασία. Αυτό το σύνθημα από μόνο το ακούγεται καλό, αλλά από την άλλη είναι λαϊκιστικό και νομίζω ότι θα οδηγήσει σε ε, πάρα πολύ δεσμευτικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Επίσης ε, για την ε, κάρτα άσκησης επαγγέλματος, την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα αν θέλετε, και εδώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς ποια είναι η χρησιμότητα. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι θα δημιουργηθεί μια νέα βάση δεδομένων των εργαζομένων πολιτών. Γιατί μόνο επί τη βάση μιας τέτοιας κάρτας δεδομένων θα είναι δυνατόν να εκδοθούν τέτοιου είδους κάρτες, τέτοιου είδους δελτία Μια τέτοια θα έλεγα τράπεζα δεδομένων θα πρέπει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης από υπηρεσίες των κρατών μελών επί τη βάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. με τις άδειε οι οποίες ανακαλούνται νομίζω ότι και αυτό θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνεται αντικείμενο διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μόνο έτσι θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ένας εργαζόμενος ο οποίος δεν έχει την άδεια άσκηση επαγγέλματο σε μια χώρα δεν θα μπορέσει να την ασκήσει, να το ασκήσει το επάγγελμά του σε μια άλλη χώρα. Συνεπώς λοιπόν, κλείνοντας θα ήθελα να πω ότι μπορεί να υπάρξει από ό,τι φαίνεται ε, σωστή συνεργασία ανάμεσά μας και έτσι θα οδηγηθούμε σε μια ικανοποιητική γνωμοδότηση για την Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και επαναλαμβάνω 14 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι θα συναντηθούμε ελπίζω με όλους τους σκιώδεις εισηγητές. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Χαρτ. Ευχαριστώ. Εκπροσωπώ σήμερα τη σκιώδη συγγήτρια την κυρία Στάιντρουκ που δεν μπορούσε να είναι παρούσα και μου ζήτησε να παρουσιάσω ορισμένα θέματα σχετικά με αυτήν την οδηγία ε, διότι η κυρία Στάιντρουκ μου είπε ότι θεωρεί ε, ότι πρέπει να υπάρχει μία κοινωνική αντιμετώπιση γι' αυτό και τονίζει ε, την συνεργασία συνεργασία με τα ε, επαγγελματικά επιμελητήρια και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κυρία Στάινμπρουκ είναι θετική ε, στο να υπάρξει μία μείωση ορισμένων επαγγελμάτων αρκεί αυτό να συμβεί σε όλους τους τομείς και όχι μόνο σε λίγους επιλεγμένους. Επίσης ε, όσον αφορά τις τροπολογίες ε, και τον εξυγχρονισμό της οδηγίας ε, χαιρετίζει ότι αυτό πρέπει να συνδυαστεί με τη διαδικασία της Μπουλόνια και το πλαίσιο των επαγγελματικών ε, προδιαγραφών και ότι ε, χρειάζεται επιμόρφωση η οποία θα πρέπει να επεκταθεί από την ισχύουσα. Ε, όσον αφορά τις γνώσεις των ατόμων στα οποία αφαιρείται η άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος θεωρεί η κυρία Στάινμπρουκ ότι αυτό είναι μια πολύ γραφειοκρατική δαπάνη και θα πρέπει να αφαιθεί στους εργοδότες και θα ήταν καλό να μπορέσει να ε, επεκταθεί το θέμα της πληροφόρησης. Επίσης όσον αφορά τις γλωσσικές εξετάσεις θεωρεί ότι η ε, γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι σημαντικό στοιχείο για την ε, ένταξη στο εργατικό δυναμικό και θεωρεί ότι ε, θα μπορεί να επιβεβαιωθεί μέσω του χρόνου φοιτήσεως. Θα πρέπει να υπάρξει στήριξη για την έκθεση αυτή, λέει η κυρία Στάινμπρουκ και προσβλέπει στην ψήφιση των τροπολογιών και στην θετική συνεργασία που θα υπάρξει εντωμεταξύ. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Χίρς. Ε, ευχαριστώ για την έκθεση. Είναι σαφές ότι είναι βασικό το θέμα αυτό για την κινητικότητα της εργασίας και γι' αυτό πρέπει να επιζητήσουμε καλύτερες ε, συνθήκες και το θέμα της επιμορφώσεως είναι σημαντικό και θα πρέπει να σκεφτούμε ε, αν ένα τέτοιο πρότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν να χρησιμοποιηθεί ρυθμιστεί επίσης για επαγγέλματα που δεν έχουν εκατότατες απαιτήσει, αλλά ε, κάποιος να μπορέσει να επικαλεστεί τις γνώσεις του για να μπορέσει να έχει πιο γρήγορα μία αναγνώριση ε, του επαγγέλματός του. Όσον αφορά τις τροπολογίες, ο αριθμός τους δείχνει ότι ε, θα υπάρξει ενεργή συζήτηση και όσον αφορά τα, τις γλωσσικές εξετάσεις είναι σαφές ότι ε, μπορεί κανείς να ε, έχει αναγνώριση των ε, επαγγελματικών του ικανοτήτων χωρίς γνώση ξένης γλώσσας αλλά θα πρέπει να, να εντάσσονται σωστά οι ανάγκες για γλωσσικές γνώσεις που να έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Δηλαδή ε, στη, Γερμανία, στη Γερμανία μπορεί κανείς ε, να τα βγάλει πέρα θαυμάσια γνωρίζοντας μόνο αγγλικά και ε, θα πρέπει να υπάρξει κάποια ευελιξία γενικότητα. Καταρχήν να μπορεί να υπάρξει αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτισης χωρίς γλωσσικές γνώσεις και μετά να προστίθενται οι γλωσσικές γνώσεις. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο τονίστηκε επίσης σχετικά με την ε, ε, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ότι χρειάζεται μία μακροχρόνια εκπαίδευση πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει ότι θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη στενότητα στα επαγγέλματα αυτά και ιδίως διότι τα συστήματα εκπαιδεύσεως στον τομέα στις διάφορες διάφορες χώρες διαφέρουν πάρα πολύ και ε, ε, ε, μπορεί σε περίπτωση που κάποιος έχει εκπαιδευτεί σε ένα διπλό σύστημα να του συνυπολογίζεται ο χρόνος φοιτήσεως σε αυτό το σύστημα και να λειτουργεί θετικά και όχι αρνητικά. Αυτές είναι οι βασικές μου παρατηρήσεις. Φαντάζομαι ότι θα συζητήσουμε συγχρόνως και για το κατά πόσο μπορεί κανείς να αφαιρέσει επαγγέλματα από αυτή τη ρύθμιση πρέπει να το ελέγξουμε και πρέπει να δούμε τι είναι εφικτό να εφαρμοστεί. Θα το δούμε στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ χαίρομαι Μίλαν διότι έκανες μία έκθεση στην οποία αντιλαμβανόμαστε ότι όλοι θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερη κινητικότητα αλλά θέλουμε να τονιστεί η σημασία της ποιότητας. Δηλαδή δεν θα υποβαθμίσουμε την ποιότητα διότι χρειαζόμαστε περισσότερο προσωπικό ανεξαρτήτως των γνώσεών τους. Πολύ σωστά λες ότι ε, θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη δομική ανεργία ε, πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτά είναι βασικά. Αλλά στη συνεδρίαση συντονισμού που παρίστασε ο Μίλαν και οι προλαλήσασες επίσης είπαμε ε, ποια είναι τα καθήκοντά μας και εγώ παραπονέθηκα ότι η έκθεση αυτή τελικώς ε, κατέληξε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ στην οποία δεν έπρεπε να βρίσκεται διότι αυτό είναι δικό μας θέμα ε, η απασχόληση μας απασχολεί εμάς και δεν είναι δυνατόν στην ΙΜΚΟ να ε, ε, μπερδεύονται παντού και οι εκθέσεις να καταλήγουν εκεί αντί για εδώ. Εδώ έχουμε πολλούς έμπειρους του τομέα και καλό θα ήταν εμείς να ξεκινούσαμε την επεξεργασία αυτής της έκθεσης η οποία είναι κατά πρωτοβουλία. Δεν καταγράφονται οπότε τη Δευτέρα μπορεί να παρουσιάσουμε μία τέτοια έκθεση μια Δευτέρα με πέντε άτομα στην αίθουσα που κανείς δεν θα ξέρει περί τίνος πρόκειται και θα παραγνωριστεί η σημασία αυτής της σημαντικής έκθεσης. Ε, Μίλαν επίσης ξέρω ότι τα γερμανικά σου είναι εξαιρετικά ε, και εγώ είπα ότι έπρεπε να προσανατολιζόμαστε σε μεγαλύτερη ποιότητα αλλά όχι μόνο για να μειώσουμε τις δυνατότητες εκπαιδεύσεως ή προσλήψεως. Θέλουμε και θέσεις εργασίας αλλά και ποιοτικές θέσεις εργασίας που να αυξάνονται κατά τρόπον ώστε ε, να μπορεί κανείς να συγκεντρώσει συγκρίνει οι ισότιμες ε, ικανότητες. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να ε, αναγνωρίζουμε ε, τα, τις επαγγελματικές ικανότητες. Θέλουμε απλώς να υπάρχουν εξετάσεις στα κράτη-μέλη που θα οδηγήσουν σε μια αναγνώριση της επαγγελματικής κατάρτασης και στο εξωτερικό. Δηλαδή τουλάχιστον στα άλλα κράτη-μέλη. Δεν ε, ε, παρκεί ε, να κοιτάζει κανείς ποιες είναι οι επαγγελματικές γνώσεις, αλλά πώς μπορούν να βελτιωθούν με τις γλωσσικές ικανότητες και άλλες. Δεν πρέπει να υπάρχει αυτόματη αναγνώριση επαγγελμάτων που δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα αναγκαία προσόντα και ε, αν δεν έχει κανείς ε, την ε, κατάρτιση θα πρέπει να μπορέσει να την καλύψει εκ των υστέρων. Όσον αφορά τις εξαιρεσει, θα πρέπει πάλι να υπάρχει μία σύγκριση να ξέρουμε εάν υπάρχουν ή όχι τα προσόντα. Είναι κάτι που θα πρέπει να γνωρίζουμε και αυτό θα πρέπει να το πούμε και στους άλλους. Διαφορετικά δεν υπάρχει ε, μία κοινή πολιτική. Αν θέλουμε να υπάρχει το ευρωπαϊκό διαβατήριο για τους νέους της Ευρώπης πρέπει να τους πούμε τι είναι τα αναγκαία προσόντα που πρέπει να έχουν και πώς θα αναγνωρίζονται τα προσόντα τους. Ε, όσον αφορά τις ε, τη γλωσσική κατάρτιση. Ε, αν δεν ξέρουμε ποιες είναι οι αναγκαίες γλώσσες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό και συμφωνώ με τις προλαλήσεις όσον αφορά τις, τη γλωσσική κατάρτιση ότι θέλει βελτίωση και πιστεύω ότι θα υπάρξει μία ενεργή συζήτηση σχετικά με την έκθεση αυτή και θα είμαι στο Στρασβούργο για να στηρίξω κατά τη συζήτηση. Ξέρεις τις απόψεις μου, δεν προσπαθώ να φρενάρω το θέμα, αλλά θα θέλαμε να υπάρχει μία δίκαιη προώθηση της ε, ε, κινητικότητας των εργαζομένων. Δεν θέλουμε ούτε να αποκλείσουμε κανέναν, ούτε να απορρίψουμε κανέναν, αλλά θέλουμε να ξέρουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί κανείς να βρει μια δουλειά. Και ε, είδα ότι στην Ισπανία παραδείγματος χάρη άκουσα ότι όσοι οι Ισπανοί νέοι λόγω της ε, καταστάσεως της χώρας είναι άνεργοι, μαθαίνουν γερμανικά γιατί στη Γερμανία τους είπαν ότι υπάρχουν ε, ανάγκες. Λοιπόν, καλό θα ήταν ε, να υπάρχει μία συζήτηση σχετικά με τις γλωσσικές ικανότητες κατά τρόπον ώστε στην Ευρώπη να αναπτυσσόμαστε όλοι μαζί και όχι να αποκλείω ένα τον άλλον. Και λυπούμε και πάλι γιατί η έκθεση αυτή ανατέθηκε στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Εδώ είναι οι αρμόδιοι και εγώ σκοπεύω να το διακηρύξω. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η τηλεόραση του Κοινοβουλίου βρίσκεται εδώ και μας, ε, μας παίρνουν για την τηλεόραση σε περίπτωση που κάποιος αναρωτιέται. Ε, οι ε, επόμενοι ομιλητές. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ έχω την τιμή να είμαι σκιώδη εκ μέρους του ΕΛΚ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας για την πολύ αξιόλογη ε, γνωμοδότησή του που είναι πολύ σημαντική για το μέλλον της οδηγίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Εκ μέρους του ΕΛΚ ε, υπέβαλα κάποιες συμπληρωματικές και το τονίζω, συμπληρωματικές τροπολογίες για να εμπλουτίσω την έκθεση, της την... την γνωμοδότηση του εισηγητού. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα αλλά θα πρέπει προηγουμένως ε, να συνταχθεί μελέτη ε, ε, κατά πόσο είναι εφικτό κάτι τέτοιο και να λάβουμε υπόψη και τα πορίσματα της διευθύνουσας ομάδας. Όπως είπε και η κυρία Χίρς, θεωρούμε ότι τα γλωσσικά τέστα θα πρέπει να γίνουν εμπόδιο στην κινητικότητα των εργαζομένων, αλλά θα πρέπει να ληφθούν ε, αυστηρότερα μέτρα και αρχές ε, για τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Εκεί οι γλωσσικέ απαιτήσει θα μπορούσαν να είναι υψηλότερε. Σε ό,τι αφορά ε, την εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και τεχνολογικά θα συμφωνούμε. Επίσης θέλουμε ε, να δώσουμε ε, κίνητρα για την κινητικότητα και θα στηρίξουμε τις ε, τροπολογίες που θα είναι υπέρ της κινητικότητας, θα βελτιώνουν τις διαδικασίες, θα μειώνουν την, τον αριθμό των κλειστών επαγγελμάτων, των ρυθμισμένων επαγγελμάτων και επίση θα διευκολύνει την αναγνώριση των προσόντων. Δεν συμφωνούμε με τροπολογίε που ζητούν εναρμόνιση του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων, γιατί θεωρούμε ότι δεν είναι ακόμη όριμη η κατάσταση, γιατί οι, συνθήκες, οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές στα κράτη-μέλη και δεν είναι όριμη η κατάσταση, ούτε δυνατή η εναρμόνιση. Επίσης, είμαστε υπέρ των καινοτόμων λύσεων, όπως ε, κοινά ευρωπαϊκά τεστ εξετάσεις γλωσσικές. θα μπορούσαμε να δούμε κατά πόσο είναι σκόπιμες κάποιες ε, τέτοιες προτάσεις ε, και αν δεν είναι υπερβολικά γραφειοκρατικές. Σε τέτοια περίπτωση δεν θα τις υποστηρίξουμε. Θα ήθελα να μας παραλάβετε, ε, κύριε Σιγητά, τις τροπολογίες που δεν θα μπορέσετε να υποστηρίξετε. Γιατί και εμείς έχουμε κάποιες αφιβολίες με ορισμένες τροπολογίες. Δεν είμαι σίγουρη ότι αντέγραψα σωστά προηγουμένως τους αριθμούς των τροπολογιών. Παρακαλώ επαναλάβετε τις. Επαναλαμβάνουμε, είμαστε υπέρ καινοτόμων λύσεων, αυτό το είπα συγγνώμη, να μην επαναλαμβάνομαι και ευελπιστώ σε αγαστή συνεργασία με τον εισηγητή, προκειμένου να συντάξουμε συμβιβαστικέ τροπολογίε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπακ, όχι κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώς να σας υπενθυμίσω γιατί είναι τόσο σημαντικό όταν αναγνωρίζονται τα επαγγελματικά προσόντα να τονίσουμε ορισμένα θέματα για να επιβεβαιώσουμε και τη συνένεσή μας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως διότι βλέπουμε τι εμπόδια αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και καταλήγουν να αναλάβουν θέσεις εργασίας ε, οι οποίες είναι κατώτερες των προσόντων τους με χειρότερη αμοιβή και αυτό οφείλεται ε, στο ότι θα, δεν υπάρχει συνένεση σχετικά με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο βαίνει ε, προς αποτυχία. Στην Αυστρία πρόσφατα ανοίξαμε τα επαγγέλματα και ε, υπήρξαν πολλές δυσάρεστες ε, ιστορίες ε, εργαζομένων που είχαν εξαιρετικές, εξαιρετικά προσόντα στις χώρες τους και χρειάστηκε να λάβουν θέσεις εργασίας οι οποίες ήταν κάτω των δυνατοτήτων τους. Η παραδείγματος χάρη διπλωματούχοι της ιατρικής για γιατροί ή ε, άτομα με ιδιαίτερες ικανότητες όπου τους ελέγχθη ότι δεν αναγνωρίστηκαν τα διπλώματά τους. Υπάρχει λοιπόν ένα τέτοιο στοιχείο. Ε, το θέμα της ποιότητος είναι πολύ σημαντικό. Η ποιότητα πρέπει να μας απασχολήσει. Αλλά εδώ μιλάμε όμως περισσότερο για διαφάνεια, για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσώνων και να μην ε, αποφεύγουμε την αναγνώριση ε, και καλυμμένα για άλλες σκοπιμότητες. Και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω μία έκκληση προς τον εισηγητή να σεβαστεί την ιδέα αυτή, ότι δηλαδή θα πρέπει να ε, αποφύγουμε ένα dumping των μισθών και να υπάρχουν πιο διάφανα μέτρα και σταθμά αξιολογήσεως ακόμη ένα θέμα. Η κυρία Σίμπελ το ανέφερα, αναφερόμαστε στους κοινωνικούς εταίρους, διότι δεν μπορούμε να τονίσουμε επαρκώς πόσο σημαντικό είναι να εμπλακούν οι κοινωνικοί εταίροι, διότι αυτοί ε, ξέρουν περί τίνος πρόκειται ε, και ποιες είναι ε, οι αναγκαίες επαγγελματικές ικανότητες για την αναγνώριση και εκεί είναι σημαντική, σημαντικό σημαντικό να εμπλακούν και οι εργοδότες αλλά και οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Έγγελ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι τροπολογίες στην έκθεση αναφέρονται σε δύο θέματα επί των οποίων πρέπει να συμφωνήσουμε. Ε, είμαι λιγάκι ενοχλημένος διότι ε, ε, θα πρέπει να τονίσω κάθε φράση του συναδέλφου Τόμας Μαν διότι δεν υπάρχει μόνο μία κρίση, μία κρίση ταυτότητα τόσα αλλά απλούστατα ε, για το γεγονός ότι ε, πρέπει να συγκλίνουν οι θέσεις μας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και θα ήθελα να τονίσω ένα θέμα το οποίο δεν τονίστηκε επαρκώς μέχρι στιγμής. Δηλαδή όποιος θέλει κινητικότητα δεν ε, μπορεί να το εξαρτήσει μονόπρευλα από την απελευθέρωση και τον, την ανταγνώριση αλλά και, την, ε, ε, και άλλους τομείς όπως οι κοινωνικές ασφαλίσεις, η κοινωνική αναγνώριση διότι διαφορετικά θα υπάρχει διάθεση ξέφρενη χωρίς όμως να λαμβάνουμε υπόψη τα κοινωνικά συμφέροντα των εργαζομένων. Εξού και πιστεύω ότι η προστασία των εργαζομένων και των καταναλωτών πρέπει εδώ να τονιστεί και να υπάρχει μία ισότιμη αντιμετώπιση των δικαιωμάτων όλων διότι εάν θέλω να αντιταχθώ εις τον εισηγητή ε, βλέπω ότι αυτός δεν μιλά για ίση αμοιβή για την ε, ίση ε, εργασία. Σε μια αλληλέγγυη Ευρώπη θα μπορεί κάποιος να δουλέψει σε μια άλλη χώρα και να αμοιβεται χαμηλότερα γιατί προέρχεται από την Ισπανία ή από μια άλλη χώρα. Δεν μπορεί αυτή να είναι η βάση επί της οποίας θα στηρίξουμε την ισότιμη αναγνώριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και τέλος, μία τελευταία παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή δεν βρέπω κανένα λόγο να μειώσουμε τα επαγγέλματα τα οποία είναι ρυθμισμένα. Αλλά θα έπρεπε να συζητήσουμε ε, για μία απλοποίηση των κανόνων αναγνωρίσεως. Γιατί ε, εγώ ξέρω από τη χώρα χώρα ότι ε, η αναγνώριση των επαγγελμάτων δεν έχει σχέση με τα επαγγελματικά προσόντα αλλά με την αντιμετώπιση των αλλοδαπών και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπερισχύσει ε, και να οδηγήσει σε επιβολή εξετάσεων και άλλων. Επίσης ε, δεν πρέπει να αποδομήσουμε ή να υποβιβάσουμε τα συστήματα ε, και να μειώσουμε τις ανάγκες και απαιτήσει επαγγελματικών προσόντων. Πρέπει να υπάρχει η καλύτερη δυνατή κατάρτιση, χρειαζόμαστε τα καλύτερα δυνατά προσόντα και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να ε, οδηγήσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους. Και τέλος ο τελευταίος ομιλητής είναι η κυρία Βίστορν και της δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ήταν ε, πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση αυτή. Πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και το είδαμε από τον μακροσκελή κατάλογο των αγορητών. Μιλούμε συνήθως για τις τέσσερις ελευθερίες, ε, ελεύθερης διακίνησης, ε, ελευθερή κυκλοφορίας προϊόντων, αγαθών, αγαθών υπηρεσιών, κεφαλαίων, αλλά νομίζω ότι έφτασε η ώρα να μιλήσουμε και για την πέμπτη ελευθερία, που θα μπορούσε να είναι η ελευθερία της γνώσης ή ελεύθερη διακίνηση της γνώσης ε, πάνω από τα εθνικά σύνορα. Φυσικά το θέμα της επαγγελματική ε, επιμόρφωσης και κατάρτισης θα πρέπει να γίνει σεβαστό και να αναγνωριστεί. Στην πατρίδα μου τη Σουηδία για δεκαετίες ολόκληρες είδαμε ότι είχαμε τους καλύτερους ταξιτζίδες και πιτσαδόρους. Ε, έχουμε και πολιτικούς μηχανικούς και ε, οδοντίατρους, αλλά εξαιτίας ε, κάποιων προκαταλήψεων ε, και μη αναγνώρισης οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να βρουν τη δουλειά που τους αξίζει. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Είναι θέμα σεβασμού τη ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και των επαγγελματικών δεξιοτήτων και των κοινωνικών δεξιοτήτων. Αυτέ θα πρέπει να γίνουν σεβαστέ σε όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί είμαστε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση κρατών μελών. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία την έγκριση της γνωμοδότησης και ευελπιστώ ότι και ο δικός μας ηγητής θα συμβάλλει στη διαμόρφωση της πολύ καλής ιδιέκθεσης ε, της ΣΥΜΚΟ. Ευχαριστώ κύριο Σκάμπρνοχ. Ε, Ευχαριστώ συνάδελφοι. Πράγματι η συζήτηση που προηγήθηκε ήταν μια πάρα πολύ πλούσια συζήτηση. Σημείωσα πάρα πολύ προσεκτικά όλα σας τα σχόλια και θα προσπαθήσω να τα εντάξω στις συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες θα προσπαθήσω να συντάξω. Όπως είπε και ο κύριος Έγγελ, για την αρχή ε, ίσης αμοιβή για την ίση εργασία, εγώ δεν την υποστηρίζω. Είναι πολύ δύσκολο Γερμανοί διαχειριστές οι οποίοι εργάζονται στη Σλοβακία σαν παράδειγμα αυτοκινητοβιομηχανίες να δεχθούν να πληρώνονται σύμφωνα με τους σλοβακικούς όρους και όχι με τους γερμανικούς όρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα τους δυσαρεστήσει ιδιαίτερα. Συνεπώς δεν δέχομαι την πρόταση αυτή. Να πω επίσης ότι δεν θα υποστηρίξω τις τροπολογίες 6 και 9. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι πάνω στο συγκεκριμένο σημείο τελειώσαμε την εξέταση των τροπολογιών. και θα κάνουμε δεκτή την έκθεση, θα την μάλλον την έκθεση αυτή στις 19 Σεπτεμβρίου. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης για την 14η οδηγία αναφέρομαι στο σημείο 12. Πρόκειται για μία γνωμοδότηση όπου εμείς πρέπει να εκφέρουμε μια γνωμοδότηση στις εργασίες της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας. Σχετικά λοιπόν με το θέμα της μεταφοράς της έδρας, εμείς πρέπει να εκφέρουμε μια γνωμοδότηση και επαναλαμβάνω ότι η αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων στις περιπτώσεις μεταφοράς της έδρας. Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να το κάνουν είναι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε αυτή την δυνατότητα για έναν μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων οι οποίες θεωρούνται περισσότερο μικρομεσαίες. Μέχρι τώρα μια οδηγία επιτρέπει τη μεταφορά της έδρας, αλλά για τις ευρωπαϊκές μόνο επιχειρήσεις και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Θα πρέπει να διευρυνθεί η δυνατότητα αυτή λοιπόν και στις υπόλοιπες επιχειρήσεις διευκολύνοντας τις μεταφορές. Σαν αντίβαρο για τη διευκόλυνση αυτή θα πρέπει εμείς να κάνουμε προτάσεις κάποιο, κάπως δεσμευτικές για την προστασία των εργαζομένων. Στόχος, εκτός από την προστασία των εργαζομένων, είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, μια πιο ολοκληρωμένη εσωτερική αγορά, στα πλαίσια πάντα της ενιαίας αγοράς. Μέσω της έκθεσής μου κάνω συγκεκριμένες προτάσεις οι οποίες επιτρέπουν την συμμετοχή των εργαζομένων στις διαδικασίες μεταφοράς. Υποχρεωτική είναι η διαβούλευση μαζί τους για το πρόγραμμα μεταφοράς με επαρκή χρονικά διαστήματα έτσι ώστε να διευκολυνθεί και να μην τους κοστίσει και κάνουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για την ίδια τη μεταφορά. Όταν υπάρχει ένα σχέδιο μεταφοράς λοιπόν το οποίο γίνεται δεκτό από τη διοίκηση και τους εκπροσώπους των εργαζομένων Εάν πράγματι οι προβλεπόμενες διατάξεις δεν εφαρμοστούν, τότε θα υπάρχει δυνατότητα νομικής προσφυγής η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στους εργαζομένους να σταματήσουν τη διαδικασία μεταφοράς ή τουλάχιστον να ζητήσουν την αναβολή της. Ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια μελέτη επιπτώσεων για την εφαρμογή αυτών των μέτρων Είδα τις 26 τροπολογίες οι οποίες κατετέθησαν, εγώ κατέθεσα 14, δεν έχω ιδιαίτερα προβλήματα με τις υπόλοιπες, νομίζω ότι συμβαδίζουμε όλοι εδώ. Κάποιες τροπολογίες είναι επακριβέστερες, είναι συμπληρωματικές και τις ε, ενσωματώνω. Για την 1, Ρέγνερ, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα. Ίσως όμως θα πρέπει να τα συζητήσουμε στα πλαίσια της οδηγίας 86-2001. Θα υπάρξουν συμβιβαστικές τροπολογίες και προτείνω στους σκιώδεις εισηγητές να συναντηθούμε στο Στρασβούργο. Έχω κάποιους μικρούς δισταγμούς σχετικά με την 26, γιατί την 26 ομολογώ δεν την καταλαβαίνω σχετικά με την δυνατότητα α, χαμηλότερου επίπεδου συμμετοχής. Λοιπόν, αυτές είναι γενικά οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Επίσης να αναφερθώ και στην τοπολογία 19 του κυρίου Άντελ ο οποίος διευκρινίζει ότι αυτό θα ισχύσει μετά την εφαρμογή της οδηγίας για την Ευρωπαϊκή Επιχείρηση. Αλλά αυτό δεν ισχύει μόνο για την λεγόμενη Ευρωπαϊκή Επιχείρηση. Νομίζω ότι θα υπάρξει συμφωνία ανάμεσά μας, θα υπάρξει συμβιβαστική προσπάθεια. Ευχαριστώ τους κοιόδης εισηγητές και όλους όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Σας ευχαριστώ. Κυρία Βίξτρομ και μετά κύριος Χέντελ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει και οδηγία εταιρικού δικαίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουλό για την ε, πολύ ισορροπημένη γνωμοδότησή του. Έχω όμως μερικές ερωτήσεις. Ε, για την τροπολογία 13, για παράδειγμα. Είπατε ότι θέλετε μία αρμόδια αρχή που θα αξιολογεί την ομότητα της μεταφοράς της έδρας εταιρεία. Θα χρησιμοποιήσουμε υπάρχουσες αρχές ή μιλάτε για τη δημιουργία μιας νέας σύσταση, μιας νέας αρμόδιας αρχής. Θα ήθελα μια διευκρίνηση. Βέβαια, εδώ βλέπουμε και τις συνέπειες πολιτικών για τις οποίες είναι αρμόδιες άλλες επιτροπές γιατί έχουμε και τη Νομική Επιτροπή και άλλες επιτροπές ε, που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Τα άρθρα 49-54 για την ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπουν ότι όλες οι εταιρείε έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε συνεπείς και η νομοθετική πρόταση που θα προκύψει να είναι ισορροπημένη γιατί ίσως να είναι νομότυπες οι μεταφορές εδρών, ακριβώς όμως επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, ίσως δημιουργηθούν κίνδυνοι για τους εργαζόμενους. Θα πρέπει να δούμε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει μια τέτοια πρόταση. Πάντως σας ευχαριστώ για την γνωμοδότηση που θα διαβάσετε στην Νομική Επιτροπή που είναι η καθήλια αρμόδια και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα ακόμη βήμα στην προσπάθεια ολοκλήρωσης εσωτερικής αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Χέντελ και μετά η κυρία Ρενή. Αγαπητοί συνάδελφοι, όταν ε, μιλάμε ε, ε, για ευρωπαϊκή ρύθμιση του δικαίου των επιχειρήσεων, του εταιρικού δικαίου θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη του την αποφυγή διευκολύσεων δηλαδή ε, που θα απευθυνθούν οι ρυθμίσεις ε, και πώς θα επηρεάσουν ε, τις ε, εθνικές αγορές. Διότι παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις ανώνυμες εταιρείες τις οποίες προτιμούν ορισμένοι από άλλες λύσεις κατά τρόπον ώστε να παραμείνουν οι αρχικές εταιρείες εν ζωή, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε μία συγχώνευση επιχειρήσεων. Οπότε πρέπει να δούμε ποια θα είναι και τα δικαιώματα των εργαζομένων που διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη στις περιπτώσεις αυτές. Ε, και πρέπει να δούμε πού θα είναι η νομική έδρα και αν μπορεί να διαχωριστεί από την διοικητική έργα και αν αυτό μπορεί να επηρεαστεί από το δικαίωμα συναποφάσεως που έχουν οι εργαζόμενοι, πράγμα το οποίο δεν είναι προφανές, διότι διαφορετικά δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι καταρτίζεται ένα νέο δίκαιο. Όσον αφορά την τροπολογία μου υπαριθμών 19, θα ήθελα να κάνω μία εξήγηση. Έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε στη συναπόφαση στη Γερμανία, δηλαδή έχουμε μία τιμή για την επόμενη φάση συναποφάσεως και στις ανώνυμες εταιρείες λέγεται ότι η κατάσταση αυτή της προηγούμενης συναποφάσεως παγώνει, πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι δεν είναι ε, σωστό και με την τροπολογία 19 θα έπρεπε ε, να υπάρχει υπάρχει το δικαίωμα επαναδιαπραγμάτευσης του τρόπου συμμετοχής που θα πρέπει να προσαρμοστεί κατά τρόπον ώστε να αυξηθούν ε, ε, ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ε, και αυτό δεν ισχύει πάντοτε. Βεβαίως εγώ εδώ αναφέρομαι ειδικά στο γερμανικό σύστημα αλλά νομίζω ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να προσταθμίσουμε, να προσαρμόσουμε στην πραγματικότητα την ισχύουσα κατάσταση και να μην αφήσουμε να περάσουν τα πάντα. Γι' αυτό και ζητώ ε, να υιοθετήσετε την τροπολογία μου 19. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι ευχαριστώ τον ε, κύριο Μπουλόν για τη συνεργασία, ε, η κυρία Ρενιέρ. ουσιαστικά έχουμε συνεργαστεί επικοδομητικά και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε έτσι. Εμείς ασχολούμαστε με την ρύθμιση των χρηματαγορών και των αναγκών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει όμως να προσέξουμε ε, διότι υπάρχει η άλλη πτυχή του εταιρικού δικαίου και δεν πρέπει εκεί να υπάρξει ξέφρενη απελευθέρωση και γι' αυτό στο θέμα της συναποφάσεως θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να καλύψουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων διότι ε, δεν διαβλέπω ποια ε, είναι η ποιος είναι ο προσανατολισμός τώρα όσον αφορά το θέμα αυτό της συναποφάσεως και θα ήθελα να μπορέσει να διευκρινιστεί διότι όταν υπάρχει μία συγχώνευση διασυνοριακή ή μία εταιρεία η οποία μεταφέρεται εκτός συνόνων, συνόρων καταστρέφεται ε, και εκεί υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν όπως είπε και ο κύριος Χέντελ δηλαδή δηλαδή ε, πρέπει να δούμε ε, ποιες θα είναι οι θεωρίες οι οποίες θα υπερισχύσουν για την εδραίωση της νέας εταιρείας και να κοιτάξουμε ε, εάν μπορούμε να βασιστούμε εις το δίκαιο για την κατάρτιση των ευρωπαϊκών εταιριών ανωνύμων εταιριών. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες αιτήσει επεμβάσεων. Πώς έχουμε κάποιον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα ήθελε να λάβει το λόγο. Ουδή. Οπότε θα ξαναδώσω το λόγο στον εισηγητή μα τον κύριο Μπουλό. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και όλου όσου ε, έλαβαν το λόγο και όσου κατέθεσαν τροπολογία στην γνωμοδότηση. Ορισμένε βέβαια ερωτήσει είναι περισσότερο νομικού χαρακτήρα και αρμόδια για τα θέματα αυτά είναι περισσότερο η νομική επιτροπή παρά η δική μας, η Επιτροπή Απασχόλησης. Πάντως, η εφαρμοστή νομοθεσία είναι η νομοθεσία της ε, χώρας υποδοχής. Αυτό προβλέπεται. Και αν η προστασία των εργαζομένων είναι ίσονη, ε, τότε εφαρμόζεται η νομοθεσία της χώρας προέλευσης, αν, είναι, ε, αν εγγυάται περισσότερα δικαιώματα. Και πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ της πραγματικής μεταφοράς και της καταστατικής μεταφοράς γιατί εδώ αναφερόμαστε στην ε, μεταφορά της καταστατικής έδρας. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξουν προβλήματα στη συνεδρία της επόμενης εβδομάδας, γιατί από ό,τι είδα υπάρχει ομόνια. Οι διαφορές αφορούν περισσότερο λεπτομέρειες ή θέματα συντακτικά. Αυτά, ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι θα ψηφίσουμε τη γνωμοδότηση αυτή στις 19 Σεπτεμβρίου ώστε να μπορέσουμε εγκαίρως να υποστηρίξουμε τη θέση μας στις 11 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Κύριε Σιγητά, πολύ συχνά υιοθετούμε εμείς τις γνωμοδοτήσεις και μετά δείχνουμε τη εμπιστοσύνη στην αρμόδια καθήλη επιτροπή. Προσοχή, εγώ είμαι στη διάθεση των εισηγητών να τους βοηθήσω και το έκανα και στο παρελθόν. Αλλά καλό είναι να δώσουμε το παρόν και στη συζήτηση στην αρμόδια καθήλη επιτροπή. Δεν είναι ότι είμαστε καχύποπτοι απέναντι στους συναδέλφους των άλλων επιτροπών, αλλά θέλουμε να είμαστε βέβαιοι ότι και οι Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτό. Νό; Νό; là, technologie me dépasse. censure. Euh... Λογοκρισία. Έτσι όταν... Μερικές φορές πέφτουμε και εμείς στην παγίδα όταν ασχολούμαστε πολύ με αυτά τα μηχανήματα. Είναι σημαντικό λοιπόν να γίνει συνάντηση και με τον συντάκτη της έκθεσης, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να επηρεάσουμε και την έκθεση. Θα έχουμε τρεις εβδομάδες με ένα μήνα, αρκετό χρόνο, αρκεί φυσικά να εγκρίνουμε μια καλή έκθεση. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό, το σημείο 12 και περνάμε στο σημείο 13 που προβλέπει εξέταση τροπολογιών για τη διαδικασία αμοιβέ αξιολόγηση τη οδηγία για τι υπηρεσίε. Συντάκτη γνωμοδότηση είναι ο κύριο Έγκελ. Έχουν κατατεθεί 21 τροπολογίε. Επί τη ουσία αρμόδια είναι η Επιτροπή ΙΜΚΟ. Αν δεν κάνω λάθο, η κυρία Μογά θα αντικαταστήσει τον κύριο Έγκελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω Συγγνώμη για τον κύριο Έγγελ που πρέπει να πάει στην Πολωνία και δεν μπορεί να πάρει το λόγο. Όπως είπατε, γι' αυτό το προσχέδιο γνωμοδότησης τη ΣΥΝΚΟ έχουν κατατεθεί 21 τροπολογίες και έχει υπάρξει μια συμβιβαστική πρόταση για τις τροπολογίες 4 και 5 για την παράγραφο 1 σχετικά με τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων απασχόλησης στις υπηρεσίες. Μια προφορική τροπολογία κανονικά θα πρέπει να παρουσιαστεί για την τροπολογία 8 της κυρίας Γκίρλινγκ. για να σβήσει μια έκφραση η οποία περιλαμβάνεται. En euh, euh, πάση περιπτώσει, ε, οι συζητήσει νομίζω ότι πήγαν πολύ καλά ανάμεσα στο σύνολο των εισηγητών και η ψηφοφορία δεν θα πρέπει να δημιουργήσει. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Τα πράγματα... Ah, alors, euh, je comprends que... Ο κύριος Σέρκας έχει ζητήσει το λόγο και με Πρώτα, πρώτα ο κύριος Σέρκας πάντως. Δεν πήρε το λόγο ο κύριος Σέρκας. Τώρα. Εν συντομία κυρία Πρόεδρε, εκ μέρους κυρίας Κίνγκα ε, που επίσης βρίσκεται εκτός Βρυξελών και δεν μπορεί να σας παρουσιάσει τη θέση των σοσιαλιστών, την αναπληρώνω εγώ, έχω τις σημειώσεις της και μου έδωσε και αρκετές πληροφορίες για να σας διαβιβάσω τη θέση των σοσιαλιστών. Κυρία Πρόεδρε, οι σοσιαλιστές είναι πρόθυμοι να κάνουν προσπάθειες ε, για την γνωμοδότηση αυτή που είναι σημαντική. Είναι σημαντική η οδηγία για τις υπηρεσίες και είναι σημαντικό να βελτιώσουμε με τη διαδικασία αυτή ένα εργαλείο από την οποία εξαρτάται ένα τομέα που δημιουργεί τι περισσότερε θέσει απασχόληση στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε προσπάθεια ώστε όλες οι χώρες να μπουν στο σωστό ρυθμό και να γνωρίσουν και οι οικονομικοί τελεστές ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες και η συμμετοχή στην εσωτερική αγορά προϋποθέτει σεβασμό των κοινωνικών διατάξεων, το δικαίωμα του καταναλωτή και ούτω καθεξής. Ο διάλογος ήταν επικοδομητικός. Αλλά δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με την έκβαση του, γιατί Καταθέσαμε τρεις μόνο τροπολογίες. Ήμασταν πολύ μετριοπαθείς λοιπόν στις αξιώσεις μας, αλλά δεν ήταν αναμενόμενη η ανταπόκριση του εισηγητού, ιδιαίτερα για τις δύο τροπολογίες, τη 14 και τη 16, για τις οποίες τουλάχιστον περιμέναμε κάποιες εξηγήσει. Γιατί δεν ε, γίνονται δεκτές. Γιατί μας λέει απλώς ότι τις απορρίπτει, αλλά δεν προτείνει καμία ε, συμβιβαστική πρόταση. Στην τροπολογία 14 απλώ λέμε ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την ανταλλαγή των πληροφοριών για θέματα που αφορά, αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και χρειαζόμαστε ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Σημαντικό να το, το τονίσουμε και η τροπολογία 16 ζητά τη διαμόρφωση ενός διαφανούς πλαισίου ώστε αυτός που παραβιάζει το νόμο να μπορεί να δώσει λόγο, να είναι υπόλογο απέναντι στους καταναλωτές για τη συμπεριφορά του. Ερωτώ λοιπόν τον εισηγητή. Ποια είναι η απάντησή του σε αυτές τις τροπολογίες. Αν διαφωνεί με τις συγκεκριμένες τροπολογίες, τι εναλλακτική λύση προτείνει. Γιατί για να υπερψηφίσουμε την έκθεση θα πρέπει να έχουμε προηγουμένως επικοδομητικό διάλογο, τουλάχιστον μια απάντηση γιατί απορρίπτονται ορισμένες θέσεις και έχουμε όλη την καλή διάθεση και την προθυμία να υπερψηφίσουμε την έκθεση. Κυρία Βίκστρομ, σας ευχαριστώ. Εγώ εκπροσωπώ τον κύριο Κρόιτσμαν που δυστυχώς απουσιάζει σήμερα. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένες παρατηρήσεις του. Έχει πολλές θέσεις και πολύ ξεκαθαρισμένες και κατηγορηματικές για την οδηγία. Ο κύριος Κρόιτσμαν κατέθεσε και τροπολογίες στη γραμμαδότηση γιατί πιστεύει ότι ε, το σχέδιο γνωμοδότηση είναι μια πολύ καλή αφετηρία για τις διαπραγματεύσεις. Η διαδικασία αμοιβέ αξιολόγηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες είναι σημαντικό εργαλείο, κατά τη γνώμη του κ. Κρότσμαν, για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς και την ε, ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης και της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, οι υπηρεσίες ε, ε, ήταν το μέσο που κατεξοχή δημιούργησε θέσεις απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τροπολογία 20 του κ. Κρόισμεντ υπογραμμίζεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κινητήριος μοχλός της ε, κοινωνικής ένταξης ε, και της απασχόλησης και δεν θα πρέπει να πλήττονται από δυσανάλογες απαιτήσει. Επίσης υπάρχει, υπηρεσιών, ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα πρέπει να αποφελούνται από τα δικαιώματά τους που πορεύουν από την εσωτερική αγορά. Γι' αυτό και ο κύριος Κρόισμαν επιδοκιμάζει την αξιολόγηση που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα τέτοιων εργαλείων. Ο κύριος Κρόισμαν συμφωνεί με την κυρία Γκέν ότι το, τα σημεία ενιαίας, ενιαίων συμβάσεων διαδραματίζουν ρόλο στην ε, οδηγία σημαντικό και η σωστή τους ε, λειτουργία θα πρέπει να αξιολογηθεί. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία 18, ο κύριος Κρόσμαν πιστεύει ότι τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα πρέπει να τύχουν προστασίας, αλλά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και τα δικαιώματα των... για τους μισθούς θα πρέπει να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό και οι φιλελεύθεροι θα ζητήσουν ξεχωριστή ψηφοφορία του συγκεκριμένου σημείου. Τέλος, ο κύριος Κρόσμαν διαφωνεί με την εισαγωγή μιας ρήτρα κοινωνική πρόοδου, όπως προτείνεται στην τροπολογία 21. Η, τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες ε, θεωρούμε ότι ήδη προστατεύονται επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Θεμελιώδων Δικαιωμάτων. Αυτά λοιπόν ήταν, ε, κυρία Πρόεδρε, τα σχόλια του κύριου Κρότσμα και τη υποφορομένης και σα ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρία Μογά, θα θέλατε να απαντήσετε εκ μέρους του εισηγητού μας. Κυρία Πρόεδρε, σημείωσα όλες τις ε, επεμβάσεις ε, θα δώσω ότι θα μεταβιβάσω τις, ε, τα σχόλια σχετικά με τις τροπολογίες αλλά καθότι δεν υπήρχε εδώ ούτε ο εισηγητής ούτε κανένα σκιώδης εισηγητής θα μπορούσαμε να έχουμε συμφωνήσει πολύ γρήγορα για τα όσα ελέγχθησαν. Εγώ όμως ε, θα μεταφέρω αυτά τα οποία ελέγχθησαν πιστότατα. Ωραία. Να επανέρχεται η συζήτηση, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να ψηφίσουμε τη Δευτέρα, διότι ελπίζω ότι μέχρι τη Δευτέρα θα μπορέσουν να επιληθούν τα προβλήματα. Ερχόμαστε τώρα στο 14 με κάποια καθυστέρηση. και ζητώ συγγνώμη διότι όσο περισσότερο χρόνο έχουμε τόσο περισσότερο σπαταλάμε. Και θα ψηφίσουμε τώρα την έκθεση Νταρντέν. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αυτό λέει η πρόεδρος το μεταφέραμε. Οπότε θα ψηφίσουμε την έκθεση 15 δηλαδή το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την εξισορρόπηση της παγκοσμιοποίησεως όπου η συγκήτρια ήταν η κυρία Χάτκιν. Σχετικά με την παράγραφο 2, τροπολογία 2, των κυρίων Σρότερ και Κορνέλισεν σε δύο μέρη. Θα ψηφίσουμε το πρώτο με μία ε, προφορική τροπολογία, δηλαδή να γράψουμε τη λέξη for και ε, χωρίς τις λέξεις prevention and. Ποιος είναι υπέρ του πρώτου αυτού μέρους υιοθετείται. Ε, ποιος είναι ε, υπέρ της διαγραφής της λέξεως end. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ξεκινά η ψηφοφορία. Ελπίζω ότι όλοι έχετε τις κάρτες σας. Κυρία Ρενιέ, έχετε την κάρτα σας. Ρέγνερ, έχετε την κάρτα σας. Λίγη ψηφοφορία. 11 υπέρ 18 κατά απερίφθη. Παράγραφος 4, τροπολογία 3 με μία προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ αυτής της τροπολογίας, κατά, αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος, αλλά νομίζω ότι απερίφθη. Ψηφίσατε όλοι. Λίγη ψηφοφορία. 10 ε, υπέρ, 18 ε, κατά, απερίφθη. Τροπολογία 4 ε, με μία προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Δεν συμφωνώ με αυτή την προφορική τροπολογία. Άρα θα ψηφίσουμε την τροπολογία 4 με την αρχική της μορφή. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μετά έχουμε ε, την τροπολογία 5. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 7, τροπολογία 6 με μία προφορική τροπολογία χωρίς αντίρρηση στην ε, προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Παράγραφος 8, τροπολογία 7 του κυρίου Ορή, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8 της κυρίας Σρότερ και Κορνέλισεν, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Παράγραφος 9, τροπολογία 9 της εισηγήτριας, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 12, τροπολογία 10 της κυρίας Χάρκιν, που θα πρέπει να τοποθετηθεί μετά την παράγραφο 6, χωρίς αντιρρήσεις, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 10, ε, μία τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μετά την παράγραφο 11, τροπολογία 12 των κυρίων Σρότερ κονέλησαν σε δύο μέρη. Ψηφίζουμε το πρώτο μέρος, Urges the Commission, ε, to Evade the Responsibilities, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο, το υπόλοιπο κείμενο, ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, μετά στην παράγραφο 11 τροπολογία 13 των ιδίων εισηγητριών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το παράγραφος 15 τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται στο εκτιμώντας 11 ε, ε, τροπολογία 1. Πρέπει να σας το εξηγήσω. Εδώ αναφερόμαστε εις ε, την εργασία της ομάδας εργασίας μας και ναι μεν ε, ε, είμαι υπέρ του, του, του, της αναγνωρίσεως της υποεπιτροπής ΦΕΜ αλλά εγώ μάλλον του Ευρωπαϊκού νομισματικού ταμείου και ε, πιστεύω ότι ουσιαστική είναι η εργασία της πλήρους επιτροπής μας και γι' αυτό και εγώ είχα προτείνει να ε, αναφέρουμε εδώ ότι είμαστε ε, στο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 Γι' αυτό εγώ πρότεινα να το διαγράψουμε αυτό, να διαγράψουμε αυτό το, το εδάφιο και ε, αυτό προτείνω, δηλαδή σας ζητώ να δεχθείτε την πρότασή μου να διαγράψουμε ε, αυτό το σημείο διότι αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι να γίνει μία προφορική τροπολογία η οποία θα λέγει αλλά θα πρέπει εδώ να αναφερθώ εις ε, τους ε, εμπειρογνώμονές μας γιατί δεν ξέρω εάν εντάχει το έχω παραβλέψει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις συζητήσεις στην Επιτροπή Απασχόλησης του The, Employment, Deliberation of the Employment Committee Ίσως να έχουμε κάποιες δυνατότητες καλύτερης ε, εξήγησης, θα έλεγα, του θέματος αυτού. Νομίζω ότι όλοι οι άλλοι συγητές θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Μα γιατί όχι, γι' αυτό σας έδωσα το λόγο και γι' αυτό θα μπορέσετε να κάνετε την παρέμβασή σας. Κοιτάξτε, η θέση μου κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα έλεγα είναι ε, δύσκολο να προσπαθεί κανείς να εκφράζει την θέση του. Εσείς το κάνετε σαν πρόεδρος και αναρωτιέμαι αν και οι υπόλοιποι συγητές έχουν την ίδια δυνατότητα. Είναι θέμα ίσων ευκαιριών. Αυτή τη δυνατότητα έχουμε πάνω σε αυτή την έκθεση η οποία είναι αρκετά σημαντική Έχουμε εργαστεί με email μόνο κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τώρα έχουμε λίγο χρόνο και έχουμε αυτή την δυνατότητα για να δώσουμε τις εξηγήσει που απαιτούνται. Αυτό συμβαίνει και σε άλλες εκθέσεις και όχι μόνο σε αυτή. Λοιπόν, η κυρία Χάρκεν, η συγγήτριά μας επί της ουσίας ουσιαστικά, έχει το λόγο. Δεν έχουμε καθόλου ήχο δυστυχώ από το μικρόφωνο της κυρίας Χάρκιν. Is that okay? Yes. Perhaps there's a message in that, anyway. Εντάξει, υπάρχει κάποιο κρυφό μήνυμα. Έχουμε καθυστερήσει την ψηφοφορία. Αυτό που άκουσα εγώ είναι είναι πιο σκληρός τρόπος ε, να διατυπώσουμε τη θέση μας. Αλλά δεν ε, είπατε ότι είναι λάθος και δεν δόθηκε καμία εξήγηση. Νομίζω ότι είναι αργά πια για να τροποποιήσουμε τον κατάλογο ψηφοφορίας. Προτιμώ να εμείνουμε σε αυτόν που έχουμε. Η πρότασή μου ήταν να τροποποιήσουμε αυτό το θεωρώντας και να ε, αναπέμψουμε το θέμα στην ε, Επιτροπή Επασχόλησης και όχι στην ομάδα εργασίας. Αν διαφωνείτε με αυτή την πρόταση, την αποσύρω και εμένουμε στην αρχική μορφή της δικής σας πρότασης. Κύριε Χάρκιν. Μήπως θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε και να αναπέμψουμε και στους δύο είναι υπερβολικό θεωρείτε. Υπάρχει αντίρρηση να ξαναστείλουμε ή μάλλον το θεωρώντας 11 να το διτυπώσουμε ως εξής. Λαμβάνοντας υπόψη τις α, α, συζητήσεις της Επιτροπής Απασχόλης και της ειδική Ομάδας Εργασίας για το Ευρωπαϊκό Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Δηλαδή να προσθέσουμε την Επιτροπή και την ειδική της ομάδα εργασίας. Κυρία Μόγα, κυρία Πρόεδρε. Βρισκόμαστε προς το τέλος ψηφοφορίας. Δεν νομίζω ότι είναι παραδεκτή μια τέτοια πρόταση. Εγώ συμμετείχα στην ομάδα Εργασίας για το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και βλέπουμε τι συμβαίνει μετά στην Ολομέλεια. Όλες οι εκθέσεις της ομάδας εργασίας που έκανε όλη την προεργασία, όλο το έργο με τις ουσίες. πάει χαμένη γιατί η Επιτροπή Απασχόλησης, ε, η Επιτροπή Συγγνώμη Προϋπολογισμού με τα οικονομικά αλλάζει τελείως ε, την ε, κατάσταση. Ουσιαστικά η Επιτροπή μας βγαίνει χαμένη απέναντι στην Επιτροπή Προπολογισμών. Καταλαβαίνω κυρία Μόρα, αλλά νομίζω ότι αυτή η πρόταση που κάνω βρίσκει σύμφωνη την Επιτροπή. Θα προσάψετε ίσως κάποια τυπολατρία, αλλά θεωρώ κάπως παράξενο, κάπως περίεργο στην Ολομέλεια να ζητάμε... Εμ, ένα σώμα που δεν είναι επίσημο σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ η Επιτροπή Απασχόληση είναι μια επίσημη επιτροπή, ένα επίσημο σώμα. Γι' αυτό είναι σημαντικό να προσθέσουμε η Επιτροπή Απασχόληση και η, η ειδικη τη ομάδα εργασία. Αν δεν υπάρχει συμφωνία, να αποσύρω την πρότασή μου. Δεν έχω αντίρρηση. Ο κύριο Ορή. ούτε κι εγώ θεωρώ σκόπιμο να κάνουμε συζήτηση εν μέσω της ψηφοφορίας. Ήδη είχαμε ένα κατάλογο ψηφοφορίας, τη θέση της ηγήτρια ας ψηφίσουμε. Άλλωστε υπάρχουν ε, σοβαρές αντιρρήσεις κατά της πρότασης. Ας ψηφίσουμε ε, ό,τι προβλέπεται στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Καλώς, αποσύρω την πρότασή μου. Και συνεχίζουμε, περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Προτιμάτε ηλεκτρονικά. Καλώς. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 27 ψήφοι υπέρ. Μία ψήφος κατά και μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Συγγετρία. Διάφορα. Αν δεν υπάρχουν, ραντεβού τη Δευτέρα του Στρασβούργου στις 7 η ώρα για την επόμενη μας συνεδρίαση.